Καλημέρα σας, αγαπητοί συνάδελφοι. Υποθέτω ότι υπάρχουν αρκετοί παρόντες σήμερα το πρωί για να μπορέσει να ξεκινήσει η συνεδρίασή μας. Καλημέρα σας. Το πρώτο μας θέμα είναι η, η υιοθέτηση του σχεδίου ημερήσιας διατάξεως που έχει κυκλοφορήσει ήδη και εάν δεν έχετε αντιρρήσεις τότε μπορούμε να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη και το δεύτερο θέμα είναι η έγκριση των πρακτικών της συνεδριάσεως 1η και 2η Σεπτεμβρίου. Εγκρίνεται επίσης και υπάρχει και η ανακοίνωση του Προέδρου ε, σχετικά με ε, τον ε, με την ε, κοινή συνεδρίαση η οποία πρόκειται να γίνεται σχετικά με την ε, συλλογική το συνολικό κανονισμό, το συλλογική απαλλαγή από τον κανονισμό των ε, αυτοκινήτων ε, στο Στρασβούργο. Θα σας πούμε πού θα γίνει, θα υπάρχει διερμηνία. Όσον αφορά την τελευταία συζήτησή μας για την ε, καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές, θα δώσω τώρα το λόγο εις ε, την εισηγήτρια κυρία Μπάρμπαρα Βάιλερ για να παρουσιάσει το ε, σχέδιο και το χρονοδιάγραμμα. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι απλούστατα μια σύντομη ανακαίνωση, ανακοίνωση διότι δεν έχω τίποτα να σας πω ο, μέχρι εκτός από την, το χρονοδιάγραμμα δηλαδή οι επόμενες ανταλλαγές επί του θέματος θα, η μία θα γίνει αύριο διότι θα έχουμε με τους σκιώδεις μία πρώτη εσωτερική ανταλλαγή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα έλεγα να συνενθούμε λίγο πιο νωρίς ε, για να μπορέσουμε να προετοιμαστούμε. Επίσης θα πρέπει να προετοιμάσουμε και την μήνυ ακρόαση για την 4η Νοεμβρίου και θα ήθελα να καλέσω όλους όσους δεν είναι σκιώδεις και ενδιαφέρονται για το φάκελο αυτό να συμβάλλουν και να διατυπώσουν προτάσεις για τα θέματα που θα ήθελαν να συζητηθούν κατά τρόπον ώστε αυτή η μήνυ ακρόαση να οργανωθεί και τα μέλη της Επιτροπής θα ενημερωθούν δηλαδή αν κάποιος έχει προτάσεις τον παρακαλώ μέχρι το τέλος της εβδομάδος να έχει υποβάλει τις προτάσεις του γιατί ε, θα, θα θα ε, καλέσουμε και την Επιτροπή Βιομηχανίας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις δημόσιες υπηρεσίες ε, οι οποίες ε, θα αναλάβουν μία νέα υποχρέωση με αυτή την ε, νέα οδηγία. Αυτές είναι οι προτάσεις μου για τους εμπειρογνώμονες και αν έχει κάποιος περαιτέρω προτάσεις μπορεί να μου τις αναφέρει αύριο το πρωί ε, στην προετοιμασία. Λοιπόν, θα κάνω στην αρχή μία παρουσίαση του εγγράφου και μετά από την ακρόαση θα καταρτήσω ένα σχέδιο εκθέσεως για να μπορέσει να είναι έτοιμο μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου και η συζήτηση θα γίνει ε, τέλος Ιανουαρίου και η ε, συζήτηση των ε, τροπολογιών για να μπορέσουμε ε, να τις συζητήσουμε και να ψηφίσουμε στην Οπτική τον Ιανουάριο και να μπορέσει να περάσει στην ε, στην ε, Ολομέλεια το Φεβρουάριο. Βλέπετε δεν είναι πολύ πιεστικό πρόγραμμα διότι ε, έχουμε συζητήσει με τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να υπάρξει αυτή η οδηγία και γι' αυτό δεν πρέπει να καθυστερήσουμε. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμά μου. Θα ήθελα να σας πω ότι δεν έχουμε ακόμη απόφαση 100% για το ποιος θα ηγηθεί, διότι η Επιτροπή διαπληκτίζεται, ε, μια άλλη Επιτροπή ε, διαπληκτίζεται με τη δικιά μας για το ποιος θα αναλάβει το θέμα αυτό αλλά το, η μεγαλύτερη πολιτική ομάδα θα έπρεπε να επέμβει διότι αν σκεφτούμε τους ενδιαφερόμενους για αυτή την ε, οδηγία που περιμένουν την νομοθεσία είναι σαφώς θέμα εσωτερικής αγοράς. Οπότε καλό θα ήταν οι συντονιστές αυτής της Επιτροπής και ε, ε, άλλοι υπεύθυνοι να συζητήσουν εις την πολιτική μας ομάδα για να διατηρήσουμε την ηγεσία αυτού του θέματος διότι το μόνο άλλο θέμα το οποίο είναι σημαντικό είναι οι νομικές πτυχές του θέματος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Βάιλερ. Υπάρχουν άλλα σχόλια, οι σκιώδεις εισηγητές μήπως θέλουν να πούν κάτι. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η σκιώδης ε, η μα μας ε, ε, δεν παρίσταται αλλά αποδίδει μεγάλη σημασία στο φάκελο αυτό διότι όπως είπατε και εσείς κυρία Βάιλερ για την εσωτερική αγορά και τις μικρές επιχειρήσεις είναι ένα πολύ βασικό θέμα που πρέπει να προωθηθεί και θα πρέπει να υπάρξει μια προστασία διότι όλες οι επιχειρήσεις δεν μεγαλώνουν υποχρεωτικά και καλό θα ήταν να μπορέσουμε να πετύχουμε. Συμφωνώ ότι το βασικό θέμα δεν είναι τα θέματα της αυτιστικής ευθύνης αλλά τα θέματα του γενικού οικονομικού πλαισίου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτό είναι κάτι το οποίο έχουμε συζητήσει ήδη ε, προτού αναλάβετε καν την έκθεση αυτή και γι' αυτό θα πρέπει η δικιά μας Επιτροπή να διατηρήσει την ηγεσία. Επίσης, ε, ο τρόπος με τον οποίο αναφέρατε ε, πώς θα διεξάγεται ε, το θέμα, συμφωνούμε. Έχω μόνο δύο προτάσεις, τις οποίες θα υποβάλω σε εσά προσωπικά μετά τη συνεδρίαση. Ευχαριστώ. Άλλα σχόλια. κύριος No. Ε, θα ήθελα να προτείνω στην κυρία Βάιλερ κατά την ε, ακρόαση να λάβουμε υπόψη και τις χώρες οι οποίες ε, πλήττονται ιδιαιτέρως ε, όπου υπάρχουν πολύ μεγαλύτερες προθεσμίες πληρωμής δηλαδή δεν είναι ε, το θέμα μόνο να συζητήσουμε για τις χώρες οι οποίες σέβονται τις προτάσεις αλλά παραδείγματο χάρη για τα νοσοκομεία σε ορισμένες χώρες η προθεσμία πληρωμής είναι 1,5 χρόνος Οπότε και αυτούς θα πρέπει να τους λάβουμε υπόψη όταν θα συζητήσουμε αυτή την οδηγία. Ο κύριος Κοτσούτσνης, θα μπορούσατε να μας πείτε πώς προφέρετε και το όνομά σας. Έντουαρτ να με λέτε. Είναι πολύ εύκολο. <laughs> Δεν είναι τόσο εύκολο, πραγματικά θέλω να ξέρω. Κοζούσνικ πρέπει να με λέτε, είναι λίγο περίπλοκο, το ξέρω. Eh, Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και θα ήθελα να σας πω ότι θα μπορέσουμε αύριο το πρωί να συμφωνήσουμε. Εγώ είμαι αναπληρωματικός και στην ε, νομική επιτροπή όπου θα συζητήσουμε σήμερα το θέμα αυτό. Οπότε και εκεί θα αφήξω τα σημεία τα οποία αναφέρατε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κουζούσνη και η κυρία Στάιλερ τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και την εισηγήτρια. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να προχωρήσουμε το θέμα των καθυστερημένων πληρωμών, διότι είναι σημαντικό θέμα, αλλά εάν είναι να γίνει ακρόαση, που από ό,τι κατάλαβα θα γίνει, είναι σημαντικό να έχουμε και εκπροσώπους από τις τοπικές κυβερνήσεις. Διότι υπάρχουν μεγάλες ανησυχίες και στις τοπικές κυβερνήσεις και πολλές τοπικές κυβερνήσεις σε διάφορες περιοχές έχουν διαφορετική εμπειρία. Στο Ηνωμένο Βασίλειο το 90% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ε, είναι, ε, των πληρωμών συγγνώμη, γίνονται καθυστερημένα και θα μπορούσαμε να δούμε και κάποιες βέλτιστες πρακτικές για το πώς ε, χρησιμοποιούνται οι διάφοροι όροι, ε, πώς μπορούμε να κάνουμε τις πληρωμές, πράγματα που μπορούμε να μάθουμε στη διάρκεια της ακρόασης. Θα ήθελα να το ζητήσω αυτό από την εισηγήτρια και επίση θα ήθελα να είμαι σαφή για το χρονοδιάγραμμα. Πολλοί από του συναδέλφου νομίζω ενδιαφέρονται για το χρονοδιάγραμμα και τι ακριβώ θα κάνουμε. Ευχαριστώ. Ο κύριο Μάγερ. Ευχαριστώ. Όσον αφορά την ιδέα του συναδέλφου Κρόιτσμαν θα ήθελα να τη συζητήσουμε ε, γιατί το έχουμε ξανασυζητήσει στο παρελθόν. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να μας παρουσιάσει έναν πίνακα για το πώς διαγράφεται η κατάσταση στα 27 κράτη-μέλη. Δηλαδή χρειαζόμαστε να έχουμε ήδη ένα σημείο συγκρίσεως. Αν έχετε τον πίνακα αυτό θα σας παρακαλούσα να μας τον δώσετε εφόσον λέτε ότι τον έχετε ήδη τον έχετε ή όχι. Όχι, ούτε η συγγήτρια δεν έχει αυτό τον πίνακα. Θα παρακαλούσα λοιπόν επισήμως να μας διανυμηθεί ο πίνακας αυτός. Να δώσω τώρα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλετε να σχολιάσετε τα όσα ακούσαμε. Mrs. Brickman. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε για το ερώτημα το οποίο ετέθη. Όντως, έχουμε διαβιβάσει μέσα στα πλαίσια της μελέτης αντικτύπου που υποβλήθηκε στην Επιτροπή σας στις αρχές Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, έχουμε διαβιβάσει τα δεδομένα, τα στοιχεία, τα οποία αφορούν τα επιμέρους κράτη-μέλη. Θα δείτε εκεί, σαφέστατα, στο κείμενο αυτό το οποίο σας διαβιβάστηκε, όλες τις πληροφορίες και όλες τις νομοθετικές ε, ρυθμίσεις που ισχύουν. Τώρα βέβαια η Κομισιό μπορεί να ε, σας παρουσιάσει συνοπτικά ξανά την, άλλη, την όλη κατάσταση, έτσι ώστε να μην υπάρχουν απορίες. Αλλά τέλος πάντων στην μελέτη αντικτύπου, στη μελέτη των συνεπειών, ούτως ή άλλως όλες αυτές τις προφορίες υπάρχουν. Πάρα πολύ ωραίο. Κυρία Μάιλερ, έχετε να κάνετε και κάποια άλλα σχόλια. Ουσιαστικά, καταλήγοντας, ευχαριστώ τους συναδέλφους για τις προτάσεις. Ε, όλοι ε, έχουμε κατακλειστεί από έγγραφα, αλλά όντως ε, είναι ένα θέμα επί του οποίου εκτός από το κείμενο λάβαμε μαζί και τον πίνακα, την ανάλυση δηλαδή, αλλά πρέπει να οργανώσουμε την ακρόαση. Είναι το πιο βασικό σημείο, διότι εκεί θα μπορέσουμε να δούμε τα βασικά θέματα της, ε, της ε, της επιφυλάξης για τις καθυστερήσεις ε, ακόμη και των πληρωμών των νοσοκομείων και εκεί θα μπορέσουμε να δούμε ε, εάν υπάρχουν ορισμένοι τομείς ε, τους οποίους δεν έχει λάβει επαρκώς υπόψη της η Επιτροπή όσο θα θέλαμε σαν Ευρωβουλευτές θα ήθελα λοιπόν να προτείνω ότι μετά από την αυριανή συζήτηση των σκιώδων εισηγητών να σηλουμε το χρονοδιάγραμμα γιατί μπορεί κάτι να προκύψει εντωμεταξύ και μετά καλό θα ήταν όλοι οι ευρωβουλευτές να έχουν το χρονοδιάγραμμα αυτό. Ευχαριστώ. Ωραία. Προς υπενθύμηση η μήνυα κρόση θα γίνει στις 4 Νοεμβρίου και ελπίζουμε να παραστούν πολλοί από τους συναδέλφους. Επόμενο σημείο στην μερίσια διάταξη. Ονομασίες και σε επισήμανση κλωστοϊφαντουργικών προϊόντων και να δώσω το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Τουάν Μάντερς, για να παρουσιάσει το χρονοδιάγραμμα και οτιδήποτε άλλο έχει να μας παρουσιάσει. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Την περασμένη εβδομάδα έγινε μια συζήτηση, μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων και αμέσως μετά έγινε μια επικοδομητική συζήτηση με τους κοιόδης συζητητές και το προσωπικό Και για να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα πρέπει να σας πω, μπορούμε απλά και μόνο να αντιγράψουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βέβαια, εμείς συμφωνήσαμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερες πληροφορίες, διότι η Επιτροπή μας είναι εσωτερική, ε, Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή και σε κάποια θέματα χρειαζόμαστε περισσότερες πληροφορίες. Το συμφώνησαν και οι σκιώδεις συγητές. Γι' αυτό και θέλουμε να τροποποιήσουμε το χρονοδιάγραμμα, όπως ακριβώς είχα προτείνει στην πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Όπως σας είπα, η συνεδρίαση με τους κοιόδης εισηγητές ήταν πολύ επικοδομητική και απέφερε καρπούς και νομίζω ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή την άγουσα γιατί την υποστήριξαν όλοι. Υπάρχουν βέβαια πολλοί που δεν συμφωνούν με την πρόταση γιατί Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που αφορούν στην προστασία του καταναλωτή, υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία υπάρχουν στο θέμα της ενημέρωσης και υπάρχει και αυτή η αξιολόγηση αντικτύπου την οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ισχυρίζεται ότι ξέρει πάρα πολλά για τα κλωστοφαντουργικά θέματα. Θα θέλουμε να έχουμε λοιπόν μία έκθεση η οποία θα την χάνει ευρεία υποστήριξη, γι' αυτό και απαιτούμε περισσότερες πληροφορίες. Να σας πω λίγο το χρονοδιάγραμμα, διότι έχουμε στην ίδια συνεδρία καθορίσει το νέο χρονοδιάγραμμα. Η αξιολόγηση αντικτύπου θα είναι έτοιμη το Δεκέμβριο, όπως προβλέπετε. Θέλουμε να γίνει μια δεύτερη ανταλλαγή απόψεων ε, κάπου στα μέσα Δεκεμβρίου Το Δεκέμβριο θα ετοιμάσω το σχέδιο έκθεσης και να το στείλω προς μετάφραση τον Ιανουάριο. Εξέταση του σχεδίου έκθεσης στα τέλη Ιανουαρίου, τροπολογίες στις αρχές Φεβρουαρίου, εξέταση τροπολογιών τέλη Φεβρουαρίου στις 23 και κατόπιν θα ψηφίσουμε ή δυνατόν στις 23 Φεβρουαρίου και πάλι στην Επιτροπή και στην ε, Ολομέλεια του Μάρτιο, ε, εάν αυτό είναι δυνατόν, τη δεύτερη Ολομέλεια του Μαρτίου του 2010. Αυτό ε, συμφωνήσαμε με τους κοιόδης εισηγητές και με το προσωπικό της γραμματείας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μάντερς. Σχόλια. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Συμφωνώ απόλυτα ότι το χρονοδιάγραμμα πρέπει να είναι πολύ ευρύτερο από αυτό που συζητήσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι, ε, θα πρέπει να έχουμε πρώτα ένα αντίγραφο της πρώτης της Κομισιόν, αλλά χρειαζόμαστε και περαιτέρω συζήτηση ε, επομένως ε, πρέπει να έχουμε στη διάθεσή μα περισσότερο χρόνο. Καλώ λέει η ε, Άλλα σχόλια. Προχωρούμε στο σημείο 6 της ημερήσιας διάταξης, ενημέρωση σχετικά με τα φάρμακα για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον εισηγητή, στον κύριο Κορέα, για να μας επιβεβαιώσει τις προθεσμίες. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει αυτή η οδηγία. Οδηγία. Όχι. Δεν είναι οδηγία. Είναι αυτός ο κανονισμός που αναφέρεται στις πληροφορίες ε, που αφορούν τον, ε, τον ασθενή και παράλληλα υπάρχει και η οδηγία η οποία συμπληρώνει την, ε, την όλη κατάσταση. Είχα ήδη ενημερώσει την Επιτροπή ΕΝΒ και νωρίτερα αλλά δεν έχω συζητήσει ακόμα με τον Κρίστοφερ ξανά. Διότι, όπως βλέπετε, και η γνωμοδότηση επί είναι από την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Γι' αυτό θα πρέπει από κοινού να ε, δούμε τις ε, δυσκολίες ε, τις οποίες παρουσιάζει το κείμενο αυτό. Πρέπει να ξέρετε ότι το κείμενο αυτό αποτελεί αντικείμενο εντόνων συζητήσεων στο Συμβούλιο, διότι υπάρχουν πάρα πολλά κράτη-μέλη τα οποία δεν συμφωνούν με την, με την πρόταση. Υπάρχουν όμως και στοιχεία τα οποία βρίσκουν σύμφωνες ε, τις ε, διάφορες αντιπροσωπίες Και, και οι δύο εισηγητές το έχουμε τονίσει αυτό. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες ε, διατάξεις οι οποίες ενισχύουν την προστασία των καταναλωτών. Και αυτές είναι διατάξεις τις οποίες δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε κατ' ουδέναν τρόπο. Δεύτερον, θα πρέπει να διευκρινίσουμε περαιτέρω όλες τις πληροφορίες οι οποίες κυκλοφορούν στο ίντερνετ και θα πρέπει να είναι και σωστές πληροφορίες, όχι πειρατικές πληροφορίες όπως ε, ε, ισχύει τώρα. Το ίντερνετ, στο ίντερνετ πρέπει να υπάρχουν σωστές επιστημονικές πληροφορίες. Και πιστεύω ότι εδώ μας προσφέρεται μια πολύ καλή ευκαιρία να έχουμε σωστές και υπεύθυνε πληροφορίες που μπορούν να αποτελέσουν και αντικείμενο καλών πρακτικών. Ε, τρίτον, με το σύνολο αυτών των κειμένων τα οποία προτίθεται και του κανονισμού και της οδηγίας που ακολουθεί ε, τονίζουμε ιδιαίτερα την προστασία. Πρέπει να προστατεύσουμε όμως περισσότερο και την προστασία του σου. Επίσης και τα δύο κείμενα και ο κανονισμός και η οδηγία δεν αλλάζουν τίποτα όσον αφορά την πληροφόρηση προς τον ε, ασθενή. Δηλαδή το, το ενημερωτικό υλικό, το ενημερωτικό φυλάδιο το οποίο υπάρχει μέσα στα φάρμακα είναι ένα κείμενο το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να το διαβάσει κανείς και να το κατανοήσει. Γι' αυτό θα πρέπει να προβλέψουμε και μια απλουστευμένη μορφή αυτού του ενημερωτικού φυλαδίου. Αυτό θα πρέπει να είναι το σημείο κίνησης για μας στο θέμα αυτό. Επίσης, πιστεύω ότι θα πρέπει να επωφεληθούμε και από τις καλές πρακτικές που ισχύουν. Παραγωγός χάρη στο σουηδικό σύστημα. Θα πρέπει να δούμε και το σουηδικό και το βρετανικό σύστημα ε, για την ε, ανέβρεση φαρμάκων. Στην Βρετανία βέβαια είναι κυρίως ε, δημόσιο το σύστημα. Στην Σουηδία είναι ένα συνδυασμός ιδιωτικού και δημοσίου συστήματος. Και οι δύο εισηγητέ ε, στην ε, γνωμοδότησή τους προτείνουν τα εξής όσον αφορά τις προθεσμίες και το χρονοδιάγραμμα. Δηλαδή 4 Νοεμβρίου παραμένει ως έχει, όσον αφορά την ε, ανάλυση της γνωμοδότησης, του σχεδίου γνωμοδότησης. Επομένως, πριν από τις 4 Νοεμβρίου δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε ακρόαση. Θεωρούμε όμως ότι μία ακρόαση είναι απολύτως απαραίτητη μετά όμως τις 4 Νοεμβρίου. Η πρώτη μερομηνία, επομένως, την οποία προτείνουμε, θα έπρεπε να αναγκάσει και τις τρεις, επιτροπή, επιτροπές να ε, επιταχύνουν τους χρόνους, ε, τους χρόνους τους. Όμως, όπως είπαμε, η ακρόαση είναι απαραίτητη. Γι' αυτό θα πρέπει να περιμένουμε να γίνει πρώτα η ακρόαση. Που δεν ξέρουμε ποια ημερομηνία θα είναι. Ίσως βέβαια θα μπορούσαμε για τις ε, τροπολογίες να επισπεύσουμε κάπως τα πράγματα. Να πούμε 11 Νοεμβρίου ε, υποβολή τροπολογιών, μετά 2 Δεκεμβρίου να συζητηθεί στην ΙΜΚΟ και 27 Ιανουαρίου στην Έμβη. Δηλαδή, είπαμε 4 Νοεμβρίου παραμένει η ημερομηνία. Κάποια στιγμή το Νοέμβριο θα γίνει μια ακρόαση μετά θα δούμε ποιο είναι το πρώτο σχέδιο γνωμοδότησης και μετά οι άλλες ημερομηνίε θα παραμείνουν όσο έχουν. Ευχαριστώ. Thank you very much, Mr. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κορέα. ο κύριος ο, ε, Μπουζόη, ο οποίος είναι ο εισηγητής στην, στο, άλλο, σχετικό κείμενο που αφορά τροποποίηση της οδηγίας, δεν έχει έρθει ακόμα. Λοιπόν, υπάρχουν σχόλια για αυτά που ακούσαμε. Όχι. Πάμε στο σημείο 8 της ημερησίας διάταξης νέες εξελίξεις σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις. Η κυρία Ρούμπλε έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Καταρχήν θα ήθελα να ε, τονίσω την ε, σημασία ε, του θέματος των δημοσίων διαγωνισμών και έχουμε ε, συζητήσει την εφαρμογή της νέας οδηγίας τελευταίως. Είχε καταρτιστεί μια έκθεση και με τον κύριο Χάμπερ Είχαμε επίσης ε, ε, συζητήσει την ανάθεση δημοσίων έργων. Με την κυρία Βάιλερ έχουμε επίσης συζητήσει μία πτυχή του θέματος και επιπλέον στην προηγούμενη νομοθετική περίοδο είχαμε καταρτήσει ακόμα ακόμη μία έκθεση. Θέλω να σας πω ότι εφόσον υπάρχει μία, ε, ένα ξεκίνημα πρέπει να συνεχιστεί διότι οι δημόσιες συμβάσεις και οι αναθέσεις τους ε, είναι, ε, ήταν ένα θέμα το οποίο τονίστηκε στην οικονομική κρίση ιδίω όσον αφορά τις κλιματολογικές αλλαγές, την χρήση διαδικασιών και προϊόντων που βλάπτουν κάπτουν το περιβάλλον και ε, είχαμε συζητήσει σε μία έκθεση και τις εμπορικές πτυχές των δημοσίων συμβάσεων διότι ε, θα πρέπει να υπάρξουν προβλέψεις για να στηριχτούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πρέπει να πω ότι ουσιαστικά ο ε, λόγος της αναθέσεως δημοσίων συμβάσεων είναι ε, για να μπορέσουν οι δημόσιες υπηρεσίες να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους και να προβούν σε αγορές με τους πλέον οικονομικούς, οικονομικά συμφέροντες όρους και προστατεύοντας το περιβάλλον και την αηφορία. Ε, δεν πρέπει να υπάρχουν όμως διακρίσεις και απαιτούμε οι διαγωνισμοί αυτοί να διευρύνουν και την εσωτερική αγορά. Αλλά ουσιαστικά το βασικό είναι να γίνεται αγορά αγαθών ε, ε, παροχής υπηρεσιών και ε, διαδικασιών που να είναι συμφέροντες. Πρέπει όμως να υπάρχει και νομική ασφάλεια με καλή, ε, με καλή παρακολούθηση και γι' αυτό πιστεύω ότι έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχουν ορισμένα ελλείμματα σε ε, ορισμένους τομείς, ε, ελλείψεις στον τομέα των κοινωνικών ε, και των περιβαλλοντολογικών και επίσης πρέπει να ξαναεξετάσουμε το ηθικό θέμα, δηλαδή το δίκαιο εμπόριο, fair trade, Υπάρχουν ορισμένες ανισορροπίες σε διάφορους τομείς, αλλά είναι δύσκολο να προβεί κανείς σε μια γενική αξιολόγηση και θα προσπαθήσω να ε, αξιολογήσω τα διάφορα στοιχεία. Το δεύτερο θέμα μας είναι η νομική ασφάλεια την ε, οποία έχουμε αναζητήσει και στο παρελθόν. Χρειαζόμαστε λοιπόν διευκρινήσεις του δικαστηρίου που είναι πολύ βασικές ε, γιατί έτσι οι infringement procedures, δηλαδή οι διαδικασίες παραβίασης θα μπορέσουν να μειωθούν στα κράτη-μέλη και υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου το οποίο επιτρέπει ή συζητά πώς πρέπει να συνεργάζονται δύο δημόσιες υπηρεσίες παραδείγματο χάρη στην περίπτωση Κομιτέλ Μπραμπάντ και σε άλλες υπάρχουν βασικές νομολογίες που λέγουν τι πρέπει να γίνεται σεβαστό στην καθημερινή εφαρμογή. Άλλωστε το, το δικαστήριο αναφέρθηκε επίσης στο θέμα των υπεργολαβιών και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη και πρέπει εδώ να πούμε ότι ε, θα υπάρχει νομική ασφάλεια και να καλέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμμορφωθεί στα συμπεφωνημένα. Καλό θα ήταν να μπορέσουμε να οργανώσουμε μία ακρόαση. Ξέρω ότι υπάρχει πίεση χρόνου, αλλά καλό θα ήταν να κάνουμε τουλάχιστον μία μίνι ακρόαση και ένα εργαστήριο διότι τα ε, δημόσια έργα αντιπροσωπεύουν 16% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα είναι ένας βασικός τομέας και γι' αυτό θα ήθελα ε, να μπορέσουμε με τους σκιώδεις συγητές να καταλήξουμε σύντομα σε μία συνεργασία και να οργανώσουμε μία πρώτη μήνυ ακρόαση. Επί του θέματος αυτά είναι τα πρώτα σχόλια που έχω. Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ ότι απαιτείται μία ακρόαση, ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη σε ένα τόσο επίκαιρο θέμα, διότι είναι μια περίοδο στην οποία θα πρέπει να επιτείνουμε τις ε, προσπάθειές μας για το κλίμα. Ο κύριος Βάρ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να σας πω ότι το ΕΛΚ στηρίζει απολύτως την πρόταση που διατύπωσε η κυρία Ρούλε και δεν έχω αυτή τη στιγμή να πω πολλά στο περιεχόμενο. Απλούστατα θα ήθελα να πω ότι δεν έχουμε καμία πίεση χρόνου. Οπότε δεν νομίζω ότι έχουμε πρόβλημα να δεν υπάρχει πρόβλημα. Μπορούμε να οργανώσουμε μία ακρόαση και με την κυρία Γκέπχαρτ και με τους συντονιστές έχουμε συζητήσει τα θέματα που είναι βασικά σε αυτήν την έκθεση. Βέβαια υπάρχουν ε, θέματα που μπορούν να βελτιωθούν, αλλά αυτό που πρέπει να εξασφαλίσουμε είναι καταρχήν να υπάρχει πλήρης διαφάνεια με ε, τις διαδικασίες και τους όρους της ε, προκήρυξης είναι διότι έτσι υπάρχει δυνατότητα να δράσει κανείς σε επίπεδο εσωτερικής αγοράς και πρέπει ε, να εφαρμόζεται και η αρχή της επικουρικότητος. Οι δημοτικές αρχές έχουν ε, ε, ελευθερία κινήσεως αλλά θα πρέπει επίσης αν ζητούν αναβολές ή παρεκκλήσεις να ελέγχονται και γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να γίνει μια σωστή συζήτηση και δεν θα πρέπει να επικαλιστούμε πρίεση χρόνου για να ε, μειωθεί αυτή η ε, έρευνα. Ευχαριστώ. Η κυρία Βάιλερ. Ε, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Ρούλε και συμφωνώ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτή η Επιτροπή να ασχοληθεί διεξοδικά με το θέμα αυτό όχι μόνο βάσει των ε, νέων αποφάσεων του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου αλλά και των προβλημάτων που προκύπτουν από τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Είναι θέμα που πρέπει να συζητηθεί διότι υπάρχουν κατ' εμάς ορισμένες αμφιλεγόμενες αποφάσεις ε, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στο παρελθόν. Δεν νομίζω δηλαδή ότι λύθηκαν όλα τα προβλήματα με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και πρέπει να το εξετάσουμε λεπτομερώς. Επίσης έχω έχω διαπιστώσει στην πρακτική ότι κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσεως η οποία ακόμη συνεχίζεται. Στην αρχή όμως ιδίω της οικονομικής κρίσεως υπάρχουν ορισμένοι εθνικοί νομοθέτες που είχα διατυπώσει ε, μία ε, απλοϊκή μορφή ε, προκηρύξεων διαγωνισμών και είναι κάτι το οποίο επίσης πρέπει να εξεταστεί ενδελεχώς να δούμε αν αυτό ήταν λογικό κατά τη διάρκεια της κρίσης και αν η σιωπηλή αποδοχή αυτών των πρακτικών ε, θα πρέπει και από την Επιτροπή μας να θεωρηθεί ότι είναι συνήθις πρακτική. Ε, αυτό ήταν το δεύτερο θέμα. Τρίτο θέμα, κυρία Ρούλε, αντιλαμβάνεστε ότι για μας ε, το ΕΛΚ, είναι, εμάς τους σοσιαλιστές είναι βασικό να εξετάσουμε τις κοινωνικές πτυχές, διότι στη Γερμανία η κατάσταση είναι ασαφής Δηλαδή υπάρχουν ε, ορισμένοι οι οποίοι προκυρήσουν διαγωνισμούς και χρησιμοποιούν τις συλλογικέ συμβάσεις και άλλοι όχι. Είναι ένα άλλο θέμα το οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψη και τέλος το τελευταίο που ανέφερε ο κύριος Σουάμπη, διαφάνεια που ακούγεται θαυμάσιο και επί σήμος κανείς ε, δημοτικός ε, σύμβουλος ή πολιτικός δεν πρόκειται να μας αντιλέξει αλλά ξέρω ότι ε, υπάρχουν ακόμη εκκρεμούσες περιπτώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και εκτός από το δίκαιο του περιβάλλοντος τα περισσότερα θέματα τα οποία εξετάζει και εκδικάζει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είναι τα θέματα των δημοσίων διαγωνισμών. Οπότε είναι, είναι αξιοπερίεργο πόσες περιπτώσεις δημοσίων διαγωνισμών καταλήγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και καλό θα ήταν να μπορέσουμε να το διευκρινίσουμε. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκέπχαρτ τώρα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ κυρία Ρούλε για την θαυμάσια σύνοψη και θα ήθελα εξ αρχής να πω για ότι συμφωνώ σε δύο θέματα τουλάχιστον, δηλαδή όντως ότι χρειάζεται μία επισκόπηση για το τι ισχύει σε αυτό τον τομέα και ε, όπου υπάρχουν αυτές οι ασαφείς καταστάσεις υπάρχει ε, κίνδυνος να υπάρχουν αμφιλεγόμενες πρακτικές και θα πρέπει να έχουμε μια σαφή εικόνα του τι ισχύει, πού και πώς και ε, πώς μπορούμε να προωθήσουμε την επίλυση. Γι' αυτό και θα ήθελα ιδίως να διαφωνήσω με ένα θέμα ε, κυρία Ρούιλε ότι έχουμε ε, πίεση χρόνου πρόκειται για μία έκθεση κατά πρωτοβουλία πρόκειται για πολύ βασικές αποφάσεις οι οποίες εξετάζονται οπότε θα πρέπει χαλαρά να μην κάνουμε μία μίνι ακρόαση αλλά μία ουσιαστική ακρόαση όπου θα ληφθούν υπόψη και τα θέματα που ανέφερε η κυρία Βάιλερ για να μπορέσουμε να ε, διατυπώσουμε ε, λέξεις, ε, λύσεις. Ένα δεύτερο θέμα επί του οποίου συμφωνώ απολύτως μαζί σας είναι ότι στο πλαίσιο αυτό πρέπει να εξετάσουμε τον ρόλο του δημοσίου. Ε, σε σχέση με τους πολίτες και δεν αναφέρομαι μόνο στην ανάθεση της σύμβασης αλλά και στο πλαίσιο μέσα στο οποίο γίνεται αυτή η ανάθεση γιατί και εσείς και η κυρία Βάιλερ είπαν ότι η κρίση απέδειξε ότι στον τομέα αυτό ε, το δημόσιο είναι ο βασικότερος ε, αναδοχός των έργων και πρέπει να δούμε λοιπόν πόσο γίνονται αυτές ε, οι ε, διακηρύξεις ε, και θα πρέπει να υπάρχει και μία νέα πτυχή νομική εις το δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων λαμβάνοντας υπόψη τα κοινωνικά κριτήρια και αν γίνονται σεβαστά ή όχι. Γιατί οι δεξιοί δεν τα επιθυμούσαν, οι αριστερά πτέρυγα το επιθυμούσε και είπαμε ότι θα δώσουμε τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν αυτές τις αρχές. Και αυτό είναι το θέμα το οποίο έθιξε τώρα η κυρία Βάιλερ, δηλαδή ότι στα κράτη-μέλη υπάρχει μία σαφής κατάσταση για το ποιος εφαρμόζει και ποιος όχι. Θα ήταν λοιπόν ίσως μία αίτηση ε, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας διευκρινίσει ποιες ε, χώρες ε, όντες εφαρμόζουν αυτά τα κριτήρια στην Ευρώπη και αυτό πρέπει να μας επηρεάσει για το πώς θα εφαρμόσουμε αυτό το κριτήριο στο μέλλον και επίσης ε, μιλώ για την πολιτική μου ομάδα συνολικά λέγοντας ότι τα κοινωνικά κριτήρια είναι πολύ βασικά και πρέπει να μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να δούμε εάν τέτοιες επιχειρήσεις ε, δεν μπορούν να προτιμηθούν εάν ε, έχουν εργαζόμενους οι οποίοι χαίρουν κοινωνικής προστασίας και κάλυψης. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ποια κριτήρια προέχουν ε, για να ασφαλίσουμε ότι υπάρχει τίμιος ανταγωνισμός και δίκαιος ανταγωνισμός μεταξύ ε, των διαγωνιζομένων ε, κατά τρόπον ώστε να μην μπορεί κανείς να αναθέτει συμβάσεις κάτω από το τραπέζι τις οποίες δεν βλέπει ο νομοθέτης. Είναι λοιπόν θέματα τα οποία πρέπει να εξετάσουμε πιο συγκεκριμένα και γι' αυτό κυρία Ρούλε σαν συντονίτρια ε, ε, είναι ίσως ένα θέμα το οποίο δεν έχει ε, συζητηθεί στην ομάδα μας αλλά σαν συντονίστρια θέλω να σας πω ότι δεν πρέπει να θεωρήσουμε ότι υπάρχει ε, χρονική πίεση και να λάβουμε όλο το χρόνο για να μπορέσουμε να ε, φωτίσουμε όλες τις πτυχές του θέματος αυτού κατά τρόπον ώστε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα χωρίς βέβαια να χρειαστεί να ε, περάσουμε δύο χρόνια αλλά εν πάση περιπτώσει δεν βιαζόμαστε και τόσο πολύ. Ευχαριστώ. Τώρα αν θα έχουμε μήνυ ακρόαση ή ολόκληρη ακρόαση θα το δούμε αυτό όταν συζητήσουμε για την, ε, το όλο χρονοδιάγραμμα. Ίσως μια πρώτη ακρόαση να είναι 1η Δεκεμβρίου. Τέλος πάντων θα το δούμε. Η κυρία Ρόιτεπε είναι η επόμενη μιλήτρια. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με όλους τους προλαλήσαντες ότι το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να εξεταστεί λεπτομερώς. Γι' αυτό και εγώ Νομίζω ότι καλό θα ήταν να υπάρξει μία πιο εκτενής ε, ακρόαση σε συνεργασία με την Περιφερειακή Επιτροπή παραδείγματος χάρη. Επίσης θα ήθελα να παρακαλέσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει ε, πού βρίσκεται η εφαρμογή της τωρινής νομοθεσίας διότι φαντάζομαι ότι όλες οι χώρες ε, προχωρούν, αλλά καλό θα ήταν να έχουμε μία επισκόπηση. Επίσης, το δεύτερο θέμα το οποίο με ενδιαφέρει είναι η κατάχρηση των ε, διαγωνισμών όπου ε, δεν γίνονται σεβαστοί οι αγώνες ανταγωνισμού και γι' αυτό θα ήθελα να παρακαλέσω την εισηγήτρια να εξετάσει και αυτή την πτυχή στην έκθεσή της και να, ε, ε, να αφιερώσει ε, ένα κεφάλαιο για να δούμε αν είναι ένα γενικό χαρακτηριστικό η παρέκκληση αυτή ή όχι. Διότι υπάρχουν δημόσιες συμβάσεις οι οποίες καταλήγουν στα δικαστήρια κατά του αναδόχου του έργου και γι' αυτό δεν πρέπει να περιορίσει κανείς το χρόνο της ε, διαπίστωσης των στοιχείων διότι έχουμε όλο και λιγότερο χρόνο υπάρχουν δηλαδή όλο και πιο συγκεκριμένες ε, προκηρύξεις διαγωνισμών και υπάρχουν συνεννοήσεις μεταξύ ε, διαφόρων συμμετεχόντων οι οποίοι συνεννοούνται μεταξύ τους όσον αφορά τις τιμές που θα προσφερθούν και πολλές φορές πριν από τον διαγωνισμό και την προκήρυξη έχει ουσιαστικά υπάρξει μία κατανομή των διαφόρων καθηκόντων. Υπάρχουν δηλαδή λανθάνοντα καρτέλ τα οποία επηρεάζουν πολύ το αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής και αυτό διαπιστώνεται και επηρεάζει την τιμή και την ποιότητα. Σε ορισμένα οικοδομικά θέματα, δρόμους ή άλλα μεγάλα τεχνικά έργα. Επίσης υπάρχει ε, ε, ε, μία ίσως τάση χώρα το, για να δούμε αν αναθέτουν σε δημόσιο οργανισμό ή σε ιδιωτικό οργανισμό το έργο αυτό. Ίσως θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάποιον τρόπο να αποκαλύψουμε αυτές τις συνεννοήσεις διότι διαφορετικά οι διαδικασίες διαγωνισμού απλώς συμβάλλουν για να συγκαλύψουν τις πρακτικές. Ευχαριστώ. Βλέπουμε και έχουμε δει και στο παρελθόν πόσο περίπλοκο είναι το θέμα αυτό διότι ίσως ε, ακόμη δεν ε, έχουμε ακόμη κοιτάξει ε, το, το θέμα της προλήψεως των ατυχημάτων. Επίσης ένα άλλο θέμα είναι η περιγραφή ε, του διαγωνισμού. Πρέπει λοιπόν να δούμε ε, πόσος χρόνος χρειάζεται για να υπάρχει νομική κάλυψη για να αποφύγει κανείς στο μέλλον ε, κάποια προσφυγή στα δικαστήρια και αυτό αναφέρεται σε προκηρύξεις μικρών δήμων ή κοινοτήτων. Γι' αυτό κυρία Ριούλε είναι πολύ σωστά όλα αυτά τα οποία είπατε. Δεν πρέπει να παρα βλέψουμε την απλοποίηση διότι δεν επιτρέπεται ε, να πρέπει κανείς να λάβει υπόψη του ατελείωτα πράγματα για να υπάρχει νομική ασφάλεια ε, για ένα ίσως επουσιώδες ε, θέμα. Δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο. Ο στόχος μας δεν είναι ε, να προσπαθήσουμε να υποχρεώσουμε τους Δήμους και τις κοινότητες να προκυρήσουν διαγωνισμούς, αλλά να διευρύνουμε την εσωτερική αγορά. Δεν πρέπει λοιπόν να ξεχνούμε ποιος είναι ο στόχος μας και ε, να διατυπώνουμε απλώς τελείωτα κριτήρια. Επίσης ένα βασικό θέμα είναι ότι ε, υπάρχουν ε, δημόσιοι οργανισμοί που αναθέτουν σε δημόσιους οργανισμούς. Οπότε τι γίνεται εκεί. Στη Γερμανία είναι πάρα πολύ βασικό το θέμα αυτό και ε, προβλέπεται σε κάποια περιοχή ότι μπορεί νομοθετικά να ανατεθεί ένα δημόσιο έργο από την ε, μία κοινότητα στην άλλη αλλά αυτό ισχύει μόνο σε δύο από τα 16 κρατήδια της Γερμανίας άρα υπάρχει ποικιλία όσον αφορά την εφαρμογή ε, των δημοσίων διαγωνισμών και συμβάσεων μην ξεχνάμε λοιπόν την απλοποίηση και την ε, διευκόλυνση των ε, άλλων. Δηλαδή ε, τι είναι τα πράγματα τα οποία επιτρέπουμε και τι πρέπει να καταλήξει στα δικαστήρια. Γιατί λοιπόν καταλήγουμε στα δικαστήρια διότι ζητούμε πάρα πολλά και τελικά οι διαδικασίες αυτές δεν είναι τόσο διάφανες. Πολύ σωστά λοιπόν είπε η συνάδελφος ότι η βασική προσπάθεια προσπάθεια της κοινότητας είναι, έχει, στόχο, ε, ε, έχει ε, στόχο να μην ξεχάσει για να μην παραβλέψει τις επιχειρήσεις της περιοχής. Υπάρχει όμως ευρωπαϊκή επιταγή η οποία απαιτεί να μην ξεχαστούν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τα δύο αυτά δεν είναι εύκολο να συνδυαστούν. Οπότε ε, πρέπει καταρχήν να δούμε ότι δεν αναθέτονται τα θέματα κάτω από το τραπέζι αλλά από την άλλη πλευρά δεν πρέπει να αγνοήσετε και τους ε, φορολογούμενούς σας, τους ε, πολίτες σας. Άρα πρέπει να υπάρχει μία ισορροπία μεταξύ όλων αυτών των θεμάτων και βλέπετε ότι ένα τεράστιο πακέτο χρειάζεται για να διατυπωθεί μία προκήρυξη διαγωνισμού ενώ θα υπαρκούσαν ίσως μερικές σελίδες. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω και ότι και εγώ συμφωνώ γιατί πρέπει να γίνει μια πλήρης ακρόαση, διότι όλοι γνωρίζουμε πώς λειτουργούν οι δημόσιες συμβάσεις στις χώρες μας, έχουμε όλοι κάποιες εμπειρίες. Και στη Σκοτία, παραδείγματος χάρη, έχουμε ένα παράδειγμα για το πώς μέσω των πολιτικών δημόσιας σύμβασης μπορέσαμε να δημιουργήσουμε ένα εργαστήρι το οποίο θα βοηθούσε τα άτομα με ειδικέ ανάγκες και τους μάθαμε εκεί για το ε, πώς ε, μπορούσαν, ε, πώς, τους μάθαμε εκεί πώς οι ευρωπαϊκές πολιτικές μπόρεσαν να τους βοηθήσουν και νομίζω ότι θα πρέπει να επωφεληθούμε όλοι από τις πρακτικές που εφαρμόζονται και ε, γι' αυτό εάν και εφόσον υπάρξει αυτή η ακρόαση να όλοι μας να παρουσιάσουμε τα παραδείγματα καλών πρακτικών και να επιλέξουμε πάρα πολύ σωστά τους συμμετέχοντες έτσι ώστε να είναι όσο το πιο συνοπτικό και, συνοπτική και σαφής η ακρόαση. Χρειάζεται λίγο χρόνο βέβαια, χρειάζεται όλο χρόνο λίγα αυτά και ευχαριστώ και την εισηγήτρια για τον τρόπο με τον οποίο μας παρουσίασε το θέμα σήμερα το πρωί. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία Ρούλε για την εισαγωγή ε, διότι όντως το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και ε, ε, θα ήθελα να το χαρακτηρίσω. Επίσης θα ήθελα να σας πω ότι από τη μία πλευρά καλό θα ήταν να ε, ελέγξουμε όλα τα θέματα και ιδίως να δούμε και τους μικρούς δήμους ε, οι οποίοι μας ρωτούν πολλές φορές μα είναι υποχρεωτικά να προκηρύξουμε ένα διαγωνισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, διότι λίγοι ούτως ή άλλως θα ενδιαφερθούν από άλλες χώρες και άρα όλη αυτή η διαδικασία δεν αξίζει τον τρόπο. Είναι κάτι που πρέπει να συζητήσουμε. Το θέμα είναι οι ο, ε, τιμές κατόφλια. Αυτό είναι το σημαντικό βέβαια ξέρω ότι η, ε, το ΕΛΚ έχει διαφορετική γνώμη από μας η Τσέσου ε, και ίσως ε, θα είναι ένα θέμα προς συζήτηση. Δεν ε, εγγυώμαι ότι θα συμφωνήσετε όλοι, αλλά είδα μία προκήρυξη αυτές τις μέρες για ένα θέμα απορριμμάτων. Μία εταιρεία ανέλαβε το έργο το, και η τοπική αρχή χρησιμοποίησε ένα κριτήριο το οποίο μετά περίφθη ε, βάσει της νομολογίας και χρειάστηκε να ξαναξεκινήσει ο διαγωνισμός ε, και ανελήφθη από κάποιον ο οποίος έδωσε μεγαλύτερη τιμή από ότι η εταιρεία της ε, περιοχής. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο πρόκειται να, πρέπει να εξετάσουμε. Επίσης τις συλλογικές συμβάσεις διότι υπάρχει διαφορά από το εάν η συλλογική ε, σύμβαση εφαρμόζεται ενιαία ή όχι και στο, το, στον τομέα των απορριμμάτων επηρεάζεται επίσης η κατάσταση από την οδηγία για τις μετακινήσεις των επιχειρήσεων και ε, όταν πρόκειται για ανθρώπους ε, και για συλλογικές συμβάσεις υπάρχουν διάφορα θέματα τα οποία είναι πολύ επίκαιρα και ε, ήθελα να παρουσιάσω αυτά τα επιχειρήματα εδώ. Ίσως μπορούμε να βρούμε έναν τρόπο να συμφωνήσουμε για το πώς θα διατυπώσουμε τις απαιτήσει μας. Ε, η πολιτική μου ομάδα ενδιαφέρει ιδιαίτερο για τις συλλογικέ συμβάσεις και θα ήθελε να περιληφθούν στα κριτήρια που θα σχολιαστούν και να δούμε επακριβώς πώς έχει η κατάσταση. Ευχαριστώ. Κάποιοι από τους συναδέλφους πρόωθησαν την ιδέα να ε, οργανώσουμε μια πλήρη ακρόαση και θα ήθελα να υπενθυμίσω στους συναδέλφους και στους συντονιστές ότι προφανώς χρειαζόμαστε κόσμο στις ακροάσεις. Πρέπει να υπάρχουν, να υπάρχουν και συμμετέχοντες. Η κυρία Μάιλερ έχει το λόγο. Με συγχωρείτε που επανέρχομαι, η κυρία Ρούλε θα καταλήξει και θα παρουσιάσει ε, τα συμπεράσματα, αλλά ε, σχετικά με τη συνάδελφο από τη Βαβαρία θα ήθελα να πω δύο πράγματα και στον κύριο Μάιερ από την ε, κάτω Σαξονία, διότι πρόσφατα είχαμε αποφασίσει μία, ένα νέο νόμο με χαμηλότερες τιμές κατόφλια και η Γερμανία ήταν από τις τελευταίες χώρες οι οποίες ε, ε, εφήρμοσαν αυτή την νομοθεσία. Θα υπήρχε λοιπόν αυτή η απλούστευση αν η Γερμανία είχε εφαρμόσει πιο νωρίς και τώρα απλώς εφαρμόζεται ένας ε, νόμος τον οποίο είχαμε συμφωνήσει προ τεσσάρων ετών και υπάρχουν νέοι δήμαρχοι οι οποίοι δεν γνωρίζουν το νέο νόμο και με λίγη εξυπνάδα καταφέρνουν να μαγειρέψουν τα αποτελέσματα. Βεβαίως ε, υπάρχουν και περιπτώσεις όπου είναι συνειδητές οι ε, ε, παρεκτροπές παρόλο που σε ορισμένες περιπτώσεις οφείλονται απλώς σε άγνοια. Και χαίρομαι που αναφέρατε το θέμα αυτό το οποίο δεν είναι όμως θέμα θέμα των, της Ευρωπαϊκής Ενώσεως αλλά των διαβουλεύσεων εις ε, το Βερολίνο. Παρακαλώ λοιπόν να ενημερώσετε εκεί τους εκπροσώπους σας. Η κυρία Ρόιτοβα ήθελε κάτι να πει ακόμη και μετά θα δώσουμε στην εισηγήτρια τη δυνατότητα να καταλήξει. Ε, τώρα θυμήθηκα κάτι, ότι ε, υπάρχει μία εφόσον υπάρχουν τόσα προβλήματα στη Γερμανία, μήπως έπρεπε η ακρόαση να γίνει στη Γερμανία Κυρία Ρότοβα μπορώ να σας πω ότι θεώρησα πολύ σημαντικά τα σχόλιά σας και όλα αυτά τα θέματα με τη, διατυπώνονται διαφορετικά στις μικρές χώρες σε σχέση με τις μεγάλες διότι ε, υπάρχει διαφορετικός τρόπος αντιμετωπίσεως στις μικρές, μεγάλες, στις μικρές χώρες και στις μεγάλες χώρες οπότε για τη δημιουργία των καρτέλ υπάρχουν θέματα που άλλοι γνωρίζουν και άλλοι όχι. Αλλά αυτό που με ενδιέφερε ήταν το θέμα των προσφυγών. Και ίσως στη Γερμανία όντως υπάρχουν εισαγγελίε οι οποίες εξειδικεύονται σε αυτές τις προσφυγές, ιδίως εφόσον υπάρχουν ασάφιες νομικές σε προκηρύξεις διαγωνισμών και νομική ανασφάλεια. Υπάρχει λοιπόν λοιπόν εδώ ε, μία ανεπάρκεια για της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διότι κοίταζε μόνο την πτυχή του δημοσίου και όχι του ιδιωτικού τομέα και οι δύο πλευρές πρέπει να λειτουργούν δίκαια και πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ε, δικαιοσύνη. Ε, ήθελα να πω και ένα άλλο θέμα το οποίο ξέχασα στην εισαγωγή. Η διαδικασία αυτή είναι πολύ σωστή και πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες, ε, πράγμα το οποίο έγινε και σχετικά με τα διαρθρωτικά ταμεία. Αλλά αυτές οι απλοποιημένες ε, διαδικασίες θα πρέπει να επιτρέπουν και διαφάνεια διότι στα πλαίσια αυτών των ε, ε, θεμάτων κατά την οικονομική κρίση είδαμε και διαφθορά και υπάρχουν ε, γκρίζες ε, περιοχές. Είναι λοιπόν κάτι που δεν πρέπει να ξεχνάμε. Πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει διαφάνεια και το πιο βασικό είναι να υπάρχει νομική ασφάλεια. Ε, γι' αυτό και καλό θα ήταν να γίνει μία συζήτηση και θα ήθελα η νομική υπηρεσία να μας στηρίξει περισσότερο σχετικά με την ανάθεση διότι έχει υπάρξει μία απόφαση στο Αμβούργο εγώ η οποία όμως πλέον δεν είναι επίκαιρη διότι διάβασα ε, γερμανικά στη μητρική μου γλώσσα τις αποφάσεις των, ε, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και πιστεύω ότι εκεί όντως δημιουργείται νομική ασφάλεια. Ευχαρίστω να σας δώσω και αγγλικές μεταφράσεις. Έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που τόσοι συνάδελφοι συμμετείχαν στη συζήτηση. Ελπίζω ότι όλοι αυτοί θα συμμετάσχουν και στην ακρόαση και ότι θα υπάρχει μια ευρία ακρόαση διότι αυτό ο, ούτως ή άλλως έχει τονιστεί ε, και από τους ε, ε, ιδιωτικούς εργολήπτες και από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και είναι ένα θέμα του οποίου ίσως οι συντονιστές θα πρέπει να αποφασίσουν. Θα ναι. ήθελα μία φράση ακόμη σχετικά με τις ε, τιμές κατόφλι. Ξέρετε ότι υπάρχει μία απόφαση ε, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, κυρία Βάιλερ, και υπάρχει νομική ανασφάλεια, διότι είχαμε ε, αποφασίσει τις τιμές κατόφλια και μετά επενέβη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ε, είχε πει ότι οι οδηγίες ισχύουν και κάτω από τις τιμές κατόφλια ε, συμφώνησε και το Κοινοβούλιο και το θέμα αυτό ακόμη δεν έχει λήξει. Άρα το επιχείρημά σας σχετικά με τις τιμές κατόφλια ε, λυπούμε αλλά δεν ισχύει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ έντονη συζήτηση. Θα περάσουμε τώρα στο επόμενο θέμα που αφορά την παρουσίαση της μελέτης με θέμα την εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Κυρία Σίλβες, μόλις ήρθε, της δίνω το λόγο. Και σας καλωσορίζω. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. θα προσπαθήσω να σας παρουσιάσω την, ε, την ομιλία μου εδώ. Έχουμε και διαφάνειες. Okay, so Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Ε, εκπροσωπώ την εταιρεία η οποία, από την οποία ζητήθηκε να συντάξει αυτή τη μελέτη σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Οι στόχοι της μελέτης ποιοι είναι. Τέσσερις βασικά. Τέσσερις στόχοι. Καταρχάς θα έπρεπε να παρουσιάσουμε μια γενική εικόνα για το, για το τι ισχύει αυτή τη στιγμή σχετικά με τη μετάθεση, εφαρμογή και ε, επιβολή της οδηγίας στα 27 κράτη-μέλη. Επίσης έπρεπε να κάνουμε μία ανάλυση των ενδεχόμενων νομικών και διοικητικών προκλήσεων που παρουσιάζει αυτή η μεταφορά σε εθνική νομοθεσία της οδηγίας. Είδαμε κάποια παραδείγματα καλών πρακτικών στα κράτη-μέλη. Και όσο σχετικά την εφαρμογή, και όσο ε, αφορά την, ε, την εφαρμογή της οδηγίας, αλλά και την εφαρμογή άλλων κανονισμών που επηρεάζουν ε, την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής της οδηγίας. Επίσης, και για να έχουμε ζωντανά παραδείγματα είδαμε και κάποιες πραγματικές ιστορίες ατόμων που συναντήσαν δυσκολίες στα διάφορα κράτη-μέλη όταν προσπαθούσαν να αναγνωρίσουν τα, τα επαγγελματικά τους προσόντα. Αυτή είναι επομένως αυτά είναι ε, ε, τα τέσσερα βασικά θέματα τα οποία θα συζητήσουμε σήμερα. Καταρχάς, α ε, ας δούμε την οδηγία αυτή καθεαυτή. Οδηγία 2005-36 ΕΚ. Η πρόταση για την οδηγία αυτή, ε, για την αναγνώριση επαγγελματικών προσώπων, ε, υποβλήθηκε μέσα στα πλαίσια της, των προτάσεων στη Σύνοδο Κορυφής της Λισαβόνας. Υιοθετήθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου του 2005 ε, ε, αποτελεί προϊόν ενοποίησης ε, πολλών προηγούμενων οδηγιών, 15 οδηγιών, ήταν 12 βασικές οδηγίες και τομεακές και τρεις οδηγίες του γενικού συστήματος. Και ομοδοποιήθηκαν όλες αυτές οι οδηγίες σε ένα και μόνο κείμενο. η βασική στόχη ήταν να ε, εξορθολογήσουμε, να πλουστεύσουμε και να βελτιώσουμε τους κανόνες για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Υπάρχουν διάφοροι στόχοι εδώ ε, για τους οποίους προσπαθήσαμε να το κάνουμε αυτό. Καταρχάς, ε, δηλαδή, να συνεισφέρουμε σε μια πιο ευέλικτη αγορά εργασίας και υπηρεσιών, να ενοποιήσουμε και να πλουστεύσουμε τα νομικά κείμενα τα οποία υπήρχαν, να βελτιώσουμε την ε, διαχείριση, την σαφήνεια και την ευελιξία, να βελτιώσουμε την ε, διοίκηση, τη διαχείριση και να βελτιώσουμε τις πληροφορίες και τις συμβουλές προς τους πολίτες και τελικά να, να καταλήξουμε σε μια απλούστερη και πιο ανοιχτή ε, κανονιστική προσέγγιση. Τώρα, τα ευρήματά μας όσον αφορά την μεταφορά και την εφαρμογή της οδηγίας. Όλα τα κράτη-μέλη, εκτός από την Ελλάδα, όλα τα κράτη-μέλη όλα τα κράτη-μέλη εκτός από την Ελλάδα έχουν μεταθέσει την οδηγία, τα 17 από τα 27 κράτη-μέλη την έχουν εφαρμόσει, πρέπει να σας πω ότι η προθεσμία για την εφαρμογή της οδηγίας είναι το 2007 δηλαδή όλα τα κράτη-μέλη έχουν καθυστερήσει, αλλά τέλο θα επανέλθουμε σε αυτό. Λόγω αυτής τη ε, καθυστερημένη ε, εφαρμογή ε, δεν μπορούμε να δούμε πώς έχει εφαρμοστεί η οδηγία, τι έχει γίνει δηλαδή και ο λόγος για τον οποίο η μεταφορά και η εφαρμογή της οδηγίας δεν σεβάστηκαν τις προθεσμίες είναι γιατί η οδηγία είναι ιδιαίτερα περίπλοκη, καλύπτει πολλούς τομείς και αρμόδιους φορείς στα κράτη-μέλη. Επίσης έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό μέτρων που πρέπει να κινητοποιηθούν εκτός από τα μέτρα τα οποία ίσχυαν μέσα στα πλαίσια των προηγούμενων τομιακών οδηγιών και η Κομισιόν ζήτησε ε, όλα τα μέτρα τα οποία έχουν υιοθετηθεί να κοινοποιηθούν ε, με βάση το άρθρο 63 της οδηγίας και αυτό σήμαινε πάρα πολύ, μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλο φόρτο εργασίας για τα κρατημέλη, εξού και οι καθυστερήσεις. Τώρα, όσον αφορά τις προκλήσεις σε προκλήσεις ε, διοικητικές ε, και νομικές. Ε, είδαμε 8 βασικές προκλήσεις. Καταρχάς το χρονοδιάγραμμα. Όπως σας είπαμε, ήταν, οι προθεσμίες δεν αρκούσαν. Κανένα κράτη-μέλη δεν μπόρεσε να εφαρμόσει, να μεταφέρει και να εφαρμόσει την οδηγία μέσα στα πλαίσια των προθεσμιών που είχαν υιοθετηθεί. Επίσης, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να δημιουργήσουμε σωστά, σωστές και ε, που να λειτουργούν σωστά δηλαδή διοικητικές δομές. Ήταν δύσκολο να γίνουν σεβαστές οι διατάξεις της οδηγίας, εξού και οι δομές που δημιουργήθηκαν δεν είναι ίδιες όλα τα κράτη-μέλη. Ε, μια άλλη πρόκληση ήταν να δημιουργήσουμε ένα απλούστερο και πλέον διαφανές σύστημα για αυτούς που διαχειρίζονται το σύστημα. Διότι, όπως σας είπα, το κείμενο είναι περίπλοκο. Προσπαθούμε να το κάνουμε απλούστερο και ε, πιο διάφανο. Παρόλα αυτά υπάρχουν πολλές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν αυτοί οι οποίοι καλούνται να διαχειριστούν το σύστημα αυτό. Επίσης, μια άλλη πρόκληση ήταν να δημιουργήσουμε μια μεγαλύτερη διαφάνεια για τους πολίτες. Αυτό έχει να κάνει και με την επικοινωνία. Επίσης, οι πολίτες δεν, ε, πρέπει, δεν μπορούν να διαβάσουν και να κατανοήσουν την οδηγία από μόνοι τους. Άρα πρέπει η, η κοινοποίηση, η ενημέρωση των πολιτών να γίνει καλύτερη. Τώρα βέβαια στα διάφορα κράτη-μέλη και η προσπάθεια διαφέρει και τα αποτελέσματα διαφέρουν. Επίσης, μια άλλη πρόκληση είναι να εξασφαλίσουμε ε, ένα σύστημα το οποίο να λειτουργεί σωστά και για τα επαγγέλματα ε, για τα οποία υπάρχει μεγάλη διασυνοριακή δραστηριότητα, ε, παραδείγματος χάρη ιατρικά επαγγέλματα, άρα και για άλλα επαγγέλματα που δεν έχουν τόσο μεγάλη διασυνοριακή δραστηριότητα. Βέβαια υπάρχει αυτό το στοιχείο του πόσο κοινό είναι το επάγγελμα, θέλετε, για το οποίο καλούνται όσοι διαχειρίζουν το σύστημα να αναγνωρίσουν τα προσόντα. Εάν έχουμε πολλά, ε, πολλούς ε, υποψήφιους από το ίδιο επάγγελμα, υπάρχει μια κάποια εξοικείωση και λειτουργούν ε, καλύτερα τα πράγματα από ό,τι για άλλα επαγγέλματα που δεν είναι τόσο συχνά. Επίσης υπάρχει μια άλλη πρόκληση που είναι η δημιουργία αμοιβαίας κατανόησης ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Και εδώ χρειάζεται να δημιουργηθεί εμπιστοσύνη ανάμεσα στα κράτη-μέλη, δηλαδή ότι ε, τα εκπαιδευτικά συστήματα καλύπτουν τα ίδια πράγματα, δηλαδή να μπορεί κάποιος να αναγνωρίζει το πτυχίο, δηλαδή όχι να, να, να θεωρεί ότι το πτυχίο ε, αντικατοπτρίζει τις ίδιες γνώσεις σε όλα τα κράτη-μέλη. Επίσης να δημιουργήσουμε μια σωστή συνεργασία ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκομένους φορείς σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, διότι είναι αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν τι συμβαίνει και στο κάτω-κάτω γνωρίζουν και τις, τα προσόντα που έχει αναποκτήσει η ενδιαφερόμενη. Επίσης θα πρέπει να εξασφαλίσουμε μια ε, προσαρμογή στις αλλαγές και μια ευελιξία στην μεταφορά. Αυτό σημαίνει ε, ότι υπάρχουν, ε, υπάρχουν πάρα πολλά, πολλές απαιτήσει ε, για τα προσόντα και τις, για τα διάφορα επαγγέλματα. Εάν μπούμε σε τόσες λεπτομέρειες όσον αφορά την περιγραφή των προσόντων και των και των, ε, και των γνώσεων, ε, κάθε φορά που αλλάζει αυτό θα πρέπει να αλλάζουμε και την νομοθεσία. Άρα οι λεπτομέρειες θα πρέπει να μπουν σε ένα παράρτημα που δεν, είναι, δεν θα είναι ε, κομμάτι του νόμου. Γιατί το παράρτημα μπορεί να προσαρμοστεί και να τροποποιηθεί συχνότερα. Και να μην χρειάζεται να αλλάζουμε και το σώμα του, του κειμένου, του νομοθετικού κειμένου. Μετά, έχουμε τις καλές πρακτικές. Τα κράτη-μέλη διαφέρουν. Άλλα κράτη-μέλη έχουν ένα ομοσπονδιακό σύστημα, όπου η οδηγία εφαρμόζεται σε ε, περιφερειακό επίπεδο, παραδείγματος στη Γερμανία και η Αυστρία, σε επίπεδο lender, Επομένως εκεί χρειάζονται μια αποκεντρωμένη προσέγγιση, ενώ άλλα κράτη-μέλη έχουν μια πιο κεντρική προσέγγιση, άρα εκεί δεν χρειάζεται συντονισμό σε περιφερειακό επίπεδο. Επίσης, εξαρτάται εξαρτάται και από τα ποια επαγγέλματα είναι κατοχυρωμένα ή είναι ρυθμισμένα, ρυθμίζονται, έχουν περιορισμούς στα κράτη-μέλη. Ε, υπάρχουν κράτη-μέλη τα οποία ρυθμίζουν και ε, προβλέπουν λεπτομέρειες για κάποια επαγγέλματα και πολλές φορές ε, ε, κάποιος επαγγελματίας δεν χρειάζεται να, να γνωρίσει κάτι όταν λειτουργεί στο δικό του, ε, στη δική του επικράτεια, ε, ενώ πρέπει να προβεί σε αναγνώριση των επαγγελματικών του προσόντων αν πρέπει να ταξιδέψει, στο, αν πρέπει να ασκήσει το επαγγελμά του στο εξωτερικό, διότι ισχύει διαφορετική νομοθεσία. Τέλο πάντων, ούτω ή άλλω θεωρούμε ότι υπάρχουν πολλέ πρακτικέ οι οποίε λειτουργούν καλά και νομίζω ότι ούτως ή άλλως και θα μπορέσουμε να αντλήσουμε διδάγματα από την εφαρμογή αυτής της οδηγίας και για, την, και για μεταγενέστερες οδηγίες. Η οδηγία για τις υπηρεσίες είναι ένα παράδειγμα ε, οδηγίας, για την εφαρμογή μιας οδηγίας δηλαδή, που είδαμε ε, ποια προβλήματα δημιούργησε και μπορέσαμε να δούμε και εδώ, να δούμε ποια προβλήματα θα μπορούσε να δημιουργήσει και αυτή η οδηγία. Πάρα πολλά κράτη-μέλη έχουν δημιουργήσει και κάποιες ε, διεπηρεσιακές ομάδες ε, που εξετάζουν την εφαρμογή της, ε, οδηγία, της μετά, μεταφορά και την εφαρμογή της οδηγίας. Αυτές οι διεπηρεσιακές επιτροπές προέρχονται από διαφορετικά υπουργεία και απαιτείται μεγάλη, ε, μεγάλος βαθμός επικοινωνίας και συνεργασίας ανάμεσα στις διάφορες υπηρεσίες των Υπουργείων. Εκεί που δημιουργήθηκε κάτι τέτοιο, αυτές οι ομάδες φαίνεται ότι βοηθούν και η κατάσταση στις χώρες αυτές είναι καλύτερη. Όχι βέβαια, αυτό δεν σημαίνει επιτάχυση της διαδικασίας, διότι πολλές φορές η ανταλλαγή περισσότερων προφοριών καθυστερεί. Αλλά τέλος πάντων, το τελικό αποτέλεσμα ήταν καλύτερο στις περιπτώσεις αυτές που υπήρχαν αυτές οι διυπηρεσιακές ομάδες. Επίσης, ε, χρειάζεται και μία συνάντηση ανάμεσα στους εθνικούς συντονιστές αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, οι συντονιστές να συναντώνται, να συζητούν, γιατί με τον τρόπο αυτό και η καθημερινή τους δουλειά γίνεται πιο εύκολη, αλλά και ε, μαθαίνουν πώς λειτουργεί το σύστημα σε άλλα κράτη-μέλη. Με τον τρόπο αυτό και το δικό τους έργο γίνεται ευκολότερο. Και ούτως ή άλλως υπάρχουν ε, δομές ε, που υπάρχουν και που λειτουργούν και θεωρούμε ότι αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή πρακτική, δηλαδή δημιουργία αυτού του δικτύου των εθνικών συντονιστών. Μετά, πρέπει να εξηγούμε και να, να ενημερώνουμε για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν, ε, λειτουργεί η νομοθεσία και σε εθνικό επίπεδο. Ε, είναι θέμα επικοινωνίας ε, δηλαδή Κάποιες χώρες έχουν ε, δημοσιεύσει ε, κάποια εγχειρίδια ή φυλάδια ενημερωτικά που βοηθούν ε, και τους διαχειριστές και αυτό είναι μια, αποτελεί μια καλή πρακτική. Επίσης κάποια εξέφρασαν την επιθυμία να δημιουργηθεί ένα template για τέτοιου είδους εγχειρίδια γιατί με τον τρόπο αυτό ε, πιστεύουμε ότι δημιουργείται και μια εναρμονισμένη προσέγγιση στα κράτη-μέλη. Και μετά υπάρχει το σύστημα, το ενημερωτικό σύστημα εσωτερικής αγοράς ε, που ε, επιτρέπει στα κράτη-μέλη να ενημερώνονται για το τι συμβαίνει το ένα στο άλλο και αυτή νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλή πρακτική διότι η ενημέρωση το τι συμβαίνει σε κάθε κράτος μέλος ε, είναι κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει και βοηθάει ιδιαίτερα. Βέβαια ε, αυτό το σύστημα δεν το χρησιμοποιούν όλα τα κράτη-μέλη στον ίδιο βαθμό, άρα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης και αυτό νομίζω η χρησιμοποίηση αυτού του συστήματος θα μπορούσε να βοηθήσει στην καλύτερη εφαρμογή της οδηγίας. We have, and you can read more about those in our report, we've looked into a number εξετάσαμε επίσης αρκετές περιπτώσεις μεμονωμένων ατόμων που προσπαθούν να αναγνωρίσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα διασυνοριακά και φυσικά οι πιο ενδιαφέρουσες περιπτώσεις είναι οι περιπτώσεις στις οποίες υπήρχαν προβλήματα. Πολλές περιπτώσεις ε, εξελίσσονται ομαλά. Αλλά είχαμε κάποιες περιπτώσεις που μας ε, δείχνουν ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα, τι προβλήματα αντιμετωπίζει κάποιος όταν προσπαθεί να εργαστεί ε, στο επάγγελμά του σε μια άλλη χώρα, ε, η οποία δεν είναι η χώρα στην οποία έλαβαν την, ε, τα επαγγελματικά αυτά προσόντα. Τα συστήματα, τα προσόντα, η μέθοδοι κατάρτισης επαγγελματιών από άλλες χώρες μέλη το γεγονός ότι είναι διαφορετικό το εκπαιδευτικό σύστημα, αυτό είναι σαφές και από τα, τα συστήματα τα ίδια και από τους ανθρώπους με τους οποίους μιλήσαμε. Τι μπορεί να κάνει λοιπόν κάποιος. Ε, η πρώτη μας σύσταση είναι ότι χρειάζεται περισσότερη επικοινωνία, περισσότερη συνεργασία και ούτω καθεξής ε, και φυσικά αυτό είναι κάτι το οποίο ελπίζουμε ότι σύντο χρόνο θα εξελιχθεί και ίσως θα έχουμε και μια πιο, θα πρέπει να υπάρχει μια πιο δραστήρια προσέγγιση για να μπορέσει να υπάρχει και μεγάλος βαθμός εμπιστοσύνης μεταξύ κρατών μελών. Ένα ουσιαστικό πρόβλημα για τους ανθρώπους που κάνουν αίτηση για αναγνώριση των προσόντων τους είναι οι καθυστερήσεις. Διότι η οδηγία λέει ότι έχουν δικαίωμα σε μια περίοδο τριών μηνών για την επίλυση της ε, ε, υπόθεσής τους, που εμείς θεωρούμε ότι είναι ένα εύλογο χρονικό διάστημα, αλλά έχουμε διαπιστώσει ότι υπήρχαν περιπτώσεις όπου χρειάστηκαν ε, χρόνια. Έχουν ε, περιπτώσει οι οποίες έχει γίνει, έχει γίνει έτσι το 2005 και ακόμα εκκρεμεί. Ε, κάποιοι δεν αναγνωρίζουν ότι υπάρχει δικαίωμα για αναγνώριση προσόντων και υπάρχει και μία τάση σε κάποια να τις καθυστερούν αυτές τις υποθέσεις για πάρα πολύ χρόνια. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι λόγω έλλειψης γνώσεων, σε κάποιες περιπτώσεις η οδηγία δεν έχει εφαρμοστεί καταλήλως και σε γενικές γραμμές δημιουργεί πολύ σοβαρά προβλήματα. Και Τέλος, σε κάποιο βαθμό υπάρχει και ένα στοιχείο προστατευτισμού, που σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη ε, ευνοούν τους ε, υπηκόους τους και δημιουργούν τεχνικά προσκόμματα για την αναχνεώρηση των ε, επαγγελματικών προσόντων. Ακόμα και αν ο τίτλο είναι λάθος, δεν αναγνωρίζουν, παρά το γεγονός ότι μιλάμε για το ίδιο επάγγελμα. Δεν αναγνωρίζουν δηλαδή αμέσω ε, ε, προσόντα από άλλο κράτος μέλος και είναι ένας τρόπος με τον οποίο προφανώς προασπίζουν τους ε, υπηκόους τους από υπηκόους άλλων κρατών μελών που έχουν τα ίδια επαγγελματικά προσόντα. Φτάνουμε λοιπόν στις συστάσεις. Να δούμε και πόσο χρόνο έχω στη διάθεσή μου. Καταρχάς λοιπόν, επειδή η οδηγία αυτή υποτίθεται ότι έπρεπε να μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο μέχρι το τέλος του 2007, έχουμε μια σημαντική καθυστέρηση. Είναι κατεπίγουσα λοιπόν η ανάγκη να διασφαλίσουμε ότι θα ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταφοράς και εφαρμογή σε όλα τα κράτη-μέλη. Κάτι το οποίο θα πρέπει να αναφέρουμε βέβαια εδώ είναι ότι ακόμα και αν κάποια κράτη-μέλη έχουν κάνει πλήρη μεταφορά και εφαρμογή της νομοθεσίας, αυτό δεν βοηθάει και πάρα πολύ εάν οι υπόλοιποι ε, δεν έχουν ε, κάνει τη μεταφορά, γιατί αυτό σημαίνει ότι το μισό σύστημα δεν λειτουργεί. Για να έχουμε λοιπόν ένα πλήρως λειτουργών σύστημα, ε, θα πρέπει να υπάρχει εφαρμογή σε όλα τα κράτη-μέλη. Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα σε αυτή την περίπτωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ε, προσφύγει στο δικαστήριο για κάποια κράτη-μέλη, αλλά φυσικά θα πρέπει να ασκηθεί και κάποια πίεση σε άλλα επίπεδα. Έχει προταθεί, για παράδειγμα, να γίνονται τακτικές συνεδριάσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Εθνικών ε, Σημείων Επαφής για να πιέσουν λίγο ε, για την ολοκλήρωση αυτή της διαδικασίας. Και αυτό που μάθαμε εδώ ήταν ότι η προθεσμία ήταν σαφέστατα πάρα πολύ φιλόδοξη. Κανένα κράτος μέλος δεν είχε ε, καταφέρει να μεταφέρει έγκαιρα. Επομένως, για το μέλλον, καλό θα ήταν Καταρχάς, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαβουλεύεται τα κράτη-μέλη και να προσπαθεί να συμφωνήσει για μια πιο εύλογη προθεσμία, Αυτό βασικά. Δηλαδή θα πρέπει να προσπαθούν να υπάρχει μια πιο εύλογη προθεσμία. Να είναι κάτι το οποίο θα είναι ρεαλιστικό ώστε η πλειονότητα των κρατών μελών τουλάχιστον να μπορούν να εφαρμόσουν την οδηγία και να τη μεταφέρουν εντό τη προθεσμία. Μετά υπάρχει το θέμα του να υπερκεράσουμε την έλλειψη εμπιστοσύνη των κρατών μελών για το σύστημα ο ένας του άλλου. Και πάλι η επικοινωνία και οι τακτικέ συνεδριάσει μεταξύ των εθνικών σημείων επαφή, το να εξοικειωθεί ο καθένα με το σύστημα ε, του άλλου για, ώστε να μπορέσουν να επιλύσουν και θέματα τα οποία μπορεί να προκύψουν, ε, είναι η σαφέστερη σύσταση που μπορούμε να δώσουμε και επίσης να επεκτείνουμε τη χρήση του ε, συστήματος IMI, ε, Internal Market Information System, και επίση υπάρχει και ένα κώδικας ε, δεοντολογίας που θα μπορούσαν να αναπτύξουν τα κράτη-μέλη. Μπορεί να μην ε, υπάρχει έλλειψη βούληση για τη χρήση αυτού του συστήματο εσωτερικών πληροφοριών, αλλά ε, μπορεί να είναι και έλλειψη ε, πόρων. Το να επισημάνουμε λοιπόν πόσο συχνά θα πρέπει να χρησιμοποιείται το σύστημα αυτό και να δημιουργήσουμε ένα καλό κώδικα διοντολογίας σημαίνει ότι θα είναι προτεραιότητα η χρήση του συστήματος σε κάποια κράτη-μέλη. Μία άλλη πρόταση είναι να εκμεταλλευτούμε την συνέργεια μεταξύ των ε, οδηγιών. Η οδηγία για τις υπηρεσίες είναι η πιο βασική σχετική υπηρεσία. Ρωτήσαμε κατά πόσον υπήρχε μια κάποια δραστηριότητα συνέργειας, ε, αν υπήρχε επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων που συμμετείχαν στη μεταφορά της μίας ή της άλλης οδηγίας στα περισσότερα κράτη-μέλη δεν υπήρχε κάτι τέτοιο φυσικά. Μια ιδέα λοιπόν θα ήταν να επιταχύνουμε αυτή την ε, συνεργασία και την επικοινωνία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, να κάνουμε τακτικές συνεδριάσεις μεταξύ των σημείων επαφής για την αναγνώριση των ε, επαγγελματικών προσόντων και των όσων είναι αρμόδιοι για την οδηγία για τις υπηρεσίες, ώστε να μπορέσουν να γνωριστούν και να συνεργάζονται μεταξύ των. Επιπλέον, σε σχέση με αυτό που μόλις είπα, κάποια κράτη-μέλη, κάποια σημεία επαφή ήταν ιδιαίτερα δραστήρια. Αρκετά από αυτά σε θέματα συνεργασίας ε, με τους εταίρους τους για την οδηγία για τις υπηρεσίες. Ίσως λοιπόν καλό θα ήταν αυτού οι οποίοι ήταν τόσο δραστηροί να συναντηθούν και να αποτελέσουν και πηγή έμπνευση ώστε να πιέσουν και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη στα οποία δεν υπάρχει τέτοια μορφή συνεργασία. Σε κάποιο βαθμό σε αρκετά κράτη-μέλη υπάρχουν ε, περιορισμοί στον προπολογισμό, γιατί φυσικά είναι αρκετή δουλειά που πρέπει να γίνει. Αυτό που θα μπορούσαμε λοιπόν να μάθουμε από τις χώρες στις οποίες ε, η συνεργασία προχώρησε ομαλά, είναι πώς να έχουμε αποτελέσματα χωρίς να πρέπει να δαπανηθούν πάρα πολλοί επιπλέον πόροι για την εφαρμογή της οδηγίας. Μετά, υπάρχει η συμμετοχή οργανώσεων του κλάδου, διότι ε, τις περισσότερες φορές οι οργανώσεις ε, του τομέα καθορίζουν τις απαιτήσεις για να μπορεί κάποιος να θεωρείται επαγγελματία στον τομέα τους. Έχουν λοιπόν πάρα πολλές γνώσεις και θα μπορούσαν να βοηθήσουν να εντοπιστούν προβλήματα και θέματα τα οποία χρήσουν επίλυσης. Υπάρχουν λοιπόν πολλές δυνατότητες οι οποίες δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ακόμα για τη συμπερίληψη των ε, ε οργανώσεων των, διαφόρων επαγγελματικών κλάδων. Ε, να ζητήσουμε για παράδειγμα ποιο είναι το συγκεκριμένο επαγγελματικό πλαίσιο προσόντων που χρειάζεται όταν, για παράδειγμα, πρέπει να εγκρίνουν ε, τα προσόντα ενός επαγγελματία από κάποιον συγκεκριμένο τομέα. Ε, σε πολύ μεγάλο βαθμό, λοιπόν, θα μπορούσαν να συνδράμουν ε, τις αρχές ώστε να μπορούν να αναγνωρίσουν τα προσόντα κάποιων και φυσικά θα δημιουργηθεί και μεγάλη εμπιστοσύνη ε, για τα συστήματα της κάθε ε, χώρας. Τέλος, Επειδή η εφαρμογή αυτή της οδηγίας υπήρξε δύσκολη και ήταν πολύ περίπλοκη διαδικασία, υπάρχει μία ανάγκη να αυξηθεί η επικοινωνία και από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει βέβαια να πω εδώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει πολλά και εκτιμάται το έργο τη από κάποια κράτη-μέλη, αλλά ε, ακόμα υπάρχει περιθώριο βελτίωση. Ε, επικοινωνία, επί μπορεί να υπάρχει με σύντομα κείμενα ή ε, μορφότυπους που εξηγούν το κείμενο της οδηγίας ή ε, επικοινωνία και με δημοσίους υπαλλήλους αλλά και με τους πολίτες καθώς επίσης και πληροφορίες για νέες αποφάσεις του δικαστηρίου ή νέες ε, ε, πληροφορίες που μπορεί να προκύψουν. Αυτά είναι μεταξύ των ετοιμάτων που λάβαμε από τα εθνικά σημεία επαφής που θα ήθελαν περισσότερη ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εν κατακλείδη, όπως σας είπα και πριν, πολλά κράτη-μέλη έχουν ήδη ετοιμάσει έγγραφα τα οποία εξηγούν με μια πιο σαφή γλώσσα πώς θα πρέπει να εφαρμόζεται η οδηγία και αυτό φυσικά θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην επικοινωνία μεταξύ των εθνικών σημείων επαφής, να υπάρχει ανταλλαγή ε, αυτών των εγγράφων καλών πρακτικών, ώστε να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν ε, και από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη και αυτά φυσικά θα γίνει ε, στις τακτικές συνεδριάσεις που γίνονται μεταξύ των σημείων επαφής. Αυτά λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις κλπ. Ευχαριστώ πολύ. Uh, Ευχαριστώ <clears throat> για αυτή την ε, παρουσίαση. Και τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα απαντήσει. Ο κύριος Γιούργεν Ντίντρε από την Γενική Διεύθυνση Αγοράς θα μας ε, σχολιάσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να σας ευχαριστήσω ιδιαιτέρως για την ευκαιρία που μου δίνετε να κάνω ορισμένες επιπλέον παρατηρήσεις σχετικά με τη μελέτη αυτή. Ίσως καλό θα ήταν να ξεκινήσω με μια προσωπική παρατήρηση. Δηλαδή ανέλαβα τη θέση αυτή από την 1η Ιουλίου. Αυτή η οδηγία είναι περίπλοκη, μου το λένε οι συνάδελφοι. Είναι μια οδηγία η οποία έχει καταρτιστεί από ειδικού για να την καταλαβαίνουν μόνο οι ειδικοί. Χαίρομαι λοιπόν ότι η η Επιτροπή σας ανέλαβε αυτή την, ε, ε, αυτό το κείμενο για να καταστεί κατανοητό και για τους κοινούς νητούς. Θα ήθελα λοιπόν να κάνω ορισμένα σχόλια και μετά να καταλήξω σε συμπεράσματα. Επειδή δηλαδή η μελέτη αυτή έγινε αγγλικά, τώρα θα περάσω στα αγγλικά. Νομίζω λοιπόν ότι η πρώτη σύσταση που έγινε στη μελέτη ήταν για να είμαστε πολύ απλοί ε, ε, διότι η περίοδος προσαρμογής που είχε αποφασιστεί ήταν πολύ περιορισμένη. Δεν θα ξανασυζητήσουμε την οδηγία τώρα, αλλά θα ήθελα να σας δώσω ορισμένες πληροφορίες όσον αφορά το περίπλοκο χαρακτήρα. Όντως ορισμένα ε, κράτη χρειάζεται να εντοπίσουν πάνω από 100 μέτρα εφαρμοστικά για αυτή την οδηγία, το οποίο είναι μεγάλη πρόκληση αλλά ε, έχουμε ξεκινήσει στην Ευρωπαϊκή Επίτροπη ε, το θέμα αυτό και βλέπουμε ότι τα κράτη-μέλη ε, αργούν να ξεκινήσουν και αρχίζουν να μας κοινοποιούν τα μέτρα που λαμβάνουν όταν εκπνέει η οδηγία αυτή. Άρα αργούν τα κράτη. Έχουμε έξι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που λέγουν, που λέγουν ότι άργησαν τα κράτη και η τελευταία απόφαση ε, ήταν αρχές Οκτωβρίου εναντίον της Γαλλίας. Ε, θα έπρεπε ίσως να κάνουμε ένα γύρο τραπέζις με τα κράτη-μέλη. Ε, είναι κάτι που κάναμε από τον Ιούνιο του 2006 και τώρα θα ήθελα να έρθω στη δεύτερη σύσταση, δηλαδή την έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ κρατών μελών για να υπερβούν τα προβλήματα. Αν κοιτάξουμε προς τα πίσω διαπιστώνουμε ότι υπήρχε μία πρόκληση μέχρι το 2004 δηλαδή ε, ε, τότε ίσχυε μία οδηγία και είχαμε δύο διευρύνσεις ε, με 12 νέα κράτη-μέλη το οποίο ήταν μεγάλη πρόκληση και επίσης από πλευράς εφαρμογής επιτόπου θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι και ο γλωσσικός φραγμός δεν είναι πουσιώδης. Άρα ε, πολύ σωστά η ε, προλαλήσασα αναφέρθηκε στο σύστημα ε, πληροφοριών και πρέπει να πω ότι είδαμε πόσες ανταλλαγές πληροφοριών έγιναν πέρυσι 1400 ετήσεις πληροφοριών ιδίως από γιατρούς και δασκάλους. 2% των ερωτήσεων αναφέρονται εις ε, ένα νέο στοιχείο που είναι η ελευθερία παροχής ε, υπηρεσιών. Ενδιαφέρον. Ε, προβλέπεται και ένας μηχανισμός σύμφωνα με τον οποίο οι εθνικοί συντονιστές μπορούν να αλλάξουν ορισμένα με ε, ε, προσαρμοστικά μέτρα. Το είπε και η προλαλή σα. Προβλέπει αυτό το ηλεκτρονικό πρότυπο την δυνατότητα να προβεί κανείς αλλαγές. Όσον αφορά τώρα την σύσταση να υπάρχουν συνέργειες με άλλες οδηγίες, το άρθρο 8 της οδηγίας υπηρεσιών θα μας απασχολήσει σε αυτό το τομέα. Ε, το τι σημαίνει είναι ότι οι ηλεκτρονικές διαδικασίες θα πρέπει να ισχύσουν και σε αυτό το τομέα και θα αρχίσει η εφαρμογή το Δεκέμβριο εφέτος. Ένα άλλο σημείο είναι ότι τα σημεία επαφής σε εθνικό επίπεδο δεν θα πρέπει να ασχοληθούν μόνο με τους συναδέλφους για την οδηγία παροχής υπηρεσιών, αλλά και ε, με ε, τα σημεία επαφής που ονομάζονται ΝΑΒΕΚ, δηλαδή ε, τους πανεπιστημιακούς ομολόγους τους. Προσπαθούμε λοιπόν να συνδυάσουμε όλες τις πτυχές και εδώ θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα θέμα. Πολύ σωστά μιλήσατε για τον ρόλο των εθνικών σημείων επαφής. Ελπίζω το Κοινοβούλιο, ε, αν ε, ε, συνεχιστεί η διαδικασία αυτή, θα τονίσει ότι πρέπει να ενταθεί συνεργασία μεταξύ των εθνικών σημείων, διότι πολλοί συνάδελφοι με ρωτούν πού είναι τα εθνικά σημεία επαφής. Αν λάβουμε υπόψη λοιπόν ότι δεν επαρκούν οι εθνικοί δεν είναι σωστή δικαιολογία για να περιμένουμε όλα να γίνουν στις Βρυξέλλες. Με συγχωρείτε που ε, τονίζω το θέμα αυτό, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, ε, η κοινωνία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τα κράτη μέλη. Τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να έρθει σε επαφή με τα κράτη-μέλη. Έχουμε συνεδριάσεις ε, ε, επιτροπών καταρτήσαμε ε, ένα μέτρο τον Ιούνιο 2009 και ε, σκοπεύουμε να, δημοσιεύσουμε άμεσα έναν οδηγό με τον οποίο σε 60 ερωτήσεις, 60 απαντήσεις θα έχετε όλες τις πληροφορίες για το τι μπορείτε να κάνετε και πώς να το κάνετε. Όσον αφορά τις οργανώσεις των διαφόρων εμπλεκομένων ε, ε, βιομηχανιών που παίζουν ένα βασικό ρόλο. Ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη εδώ το άρθρο 15 της οδηγίας για την κοινή πλατφόρμα και κατ' εμέ είναι ένα θέμα που πρέπει να δει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι είναι ένα σύστημα που δεν λειτουργεί σωστά, δεν γίνεται σωστά αντιληπτό από τις οι υπηρεσίες ε, πολλοί θεωρούν ότι είναι πολύ δύσκολο και δεν μπορεί να εφαρμοστεί άρα πρέπει να το αναθεωρήσουμε. Όσον αφορά την εμπλοκή των οργανώσεων ε, έχουμε το θέμα της επαγγελματικής κάρτας και εδώ ε, θέλω να αναφέρω ένα πρόγραμμα, μία επαγγελματική κάρτα για τους εργαζομένους στον τομέα της υγείας. Είναι άλλωστε ένα πρόγραμμα του Κοινοβουλίου και είναι το μόνο ευίωνο πρόγραμμα που έχω να υποβάλω. Συνοψίζοντας λοιπόν πιστεύω ότι η Επιτροπή έχει ασχοληθεί με το θέμα αυτό που είναι βασικό για τους πολίτες και δεν αφήνει τα πάντα απλούστατα στους εμπειρογνώμονες. Υπάρχει και ένα άγνωστο σχή στον τομέα αυτό ε, όσον αφορά τις προσωρινές παροχές υπηρεσιών και εδώ πρέπει να σας πω ότι δεν υπάρχουν επαρκή σε ανταλλαγές πληροφοριών. Υπάρχει όμως μία δυνατότητα και η δεύτερη παρατήρηση που θα ήθελα να κάνω είναι η έλλειψη, για την έλλειψη εμπιστοσύνης και πιστεύω ότι ένα στοιχείο δεν υπάρχει στη μελέτη αυτή ε, ε, ότι εξετάζουμε και άλλους τομείς και χρειάζεται να υπάρχει δικτύωση μεταξύ των αρμοδίων αρχών για τους αρχιτέκτονες, για τους επαγγελματίες θα έπρεπε να συναντούν δύο-τρεις φορές το χρόνο. Είναι κάτι που ξεκινά, αλλά εάν ε, δείτε τις αρχές ε, για τον ανταγωνισμό και προστασία των καταναλωτών τώρα πρέπει να, τώρα αρχίζουν να κινητοποιούνται ε, όταν δηλαδή παρουσιαστούν τα προβλήματα και για το μέλλον πιστεύω ότι καλό θα ήταν να ε, ε, ε, κινητοποιηθούμε περισσότερο. Δεν θα αναφερθώ στην αξιολόγηση, θα χρειαστεί να δούμε το 2020 που βρισκόμαστε, που θα είναι οι δημογραφικές εξελίξεις, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό ήταν από τα θέματα προς συζήτηση σήμερα και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έχουμε πολλούς συναδέλφου τώρα που θέλουν να μιλήσουν This topic and I now read the list. για το θέμα. Να σας διαβάσω τον κατάλογο ώστε να ξέρετε και να ελέγξετε ότι είστε στον κατάλογο. Mrs. Parvanova, then Mrs. Roitova, then Mr. Juvin, Mrs. Weiler, Mr. Lechner, Mrs. Rapti. Okay, now we start with... Ωραία λοιπόν. και ο κύριος Κέλλιν στην κατάλογο. Να ξεκινήσουμε με την κυρία Παρβάνοβα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και για την παρουσίαση η οποία νομίζω ότι έρχεται στην κατάλληλη στιγμή. Θα ήθελα να θέσω ένα θέμα το οποίο αφορά την κινητικότητα των επαγγελματιών στον τομέα της υγείας. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε το ετήσιο ε, συνέδριο το European Health Forum στη Γάσνα και μία ε, ημέρα αφιερώθηκε ιδιαίτερα στην κινητικότητα των επαγγελματιών στον τομέα της υγείας. Διότι όπως αναφέρθηκε στην παρουσίαση υπάρχει προστατευτισμός και υπάρχουν πολλά κράτη-μέλη που προσπαθούν να καθορίσουν συγκεκριμένους κανόνες που θα ε, καθυστερούν την κινητικότητα των ε, επαγγελματιών στον τομέα της υγείας και κυρίως τα σχετικά συνδικάτα σε κάθε χώρα. Υπάρχουν βέβαια κάποια τα οποία εντός εισαγωγικών θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε πιο ανεπτυγμένα κρατημέλη και εκεί υπάρχει το σύστημα των ε, επιχειρήσεων ε, ε, κυνηγών κεφαλών που ουσιαστικά παίρνουν επαγγελματίες από τα φτωχότερα Και ως επίπτωση αυτού υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις τις οποίες υπάρχουν νοσοκομεία και ιατρικά κέντρα τα οποία κλείνουν. Ε, κυρίως αφορά στις νοσοκόμες, σε κάποιες ε, χώρες ε, οι νοσοκόμες που φεύγουν από μια χώρα για να πάνε σε άλλες είναι πάνω των 10.000. Να σας δώσω το παράδειγμα της Ένωσης ε, Βουλγάρων Νοσοκόμων. Είχαμε πάρα πολλές εγγεγραμμένες, αυτή τη στιγμή είχαμε πάνω από 60.000 νοσοκόμες, αυτή τη στιγμή έχουμε λιγότερες από 30.000. Οι υπόλοιπε έχουν εξαφανιστεί από τη χώρα. Σε άλλες χώρες μελής έχουμε ελάχιστους παθολόγους και αναισθησιολόγους. Και καμιά ε, ντουζίνα παιδιάτρους. Ε, το θέμα αυτό είναι ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό το ζήτημα. Το παρουσίασαν και οι ιατρικές αρχές και οι εθνικές αρχές και αφορά το θέμα της κινητικότητας των επαγγελματιών στον τομέα της υγείας και μπορεί να φτάσουμε σε ένα στάδιο στο οποίο η ελεύθερη μετακίνηση των επαγγελματών, το οποίο σαφώ θεωρούμε βασικό ανθρώπινο δικαίωμα και συνάδει πλήρως με τα όσα ε, προσυπογράφει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτό μπορεί να ε, δημιουργήσει πολύ σοβαρό πρόβλημα να δημιουργήσει ανισότητες στον τομέα της υγείας και να αποτελέσει και σοβαρό κίνδυνο για το σύστημα υγείας. Θα παρουσιάσω και σχετική προφορική ερώτηση, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να γνωρίζουμε λίγο περισσότερο ποιες είναι οι προθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κατά πόσον ε, σκοπεύετε να κάνετε μία έρευνα, μία μελέτη, την οποία θα μπορέσετε να τη χρηματοδοτήσετε από την αξιολόγηση αντικτύπων για τους επαγγελματίες στον τομέα της υγείας και την ελεύθερη μετακίνησή τους και ποιες δράσεις ε, θα μπορούσαν να προτείνουν, διότι αυτή η μετακίνηση έχει πλέον και κοινωνικο-οικονομικές ε, επιπτώσεις. Οι κυβερνήσεις διαμαρτύρονται ότι δαπανούν πολλά χρήματα και δεν έχουν κάποιους επαγγελματίες ούτε σε ένα ούτε σε πέντε χρόνια. Είναι μεγάλη η δαπάνη και πολλά συστήματα υπάρχει περίπτωση να αντιμετωπίσουν πολύ σοβαρές δυσκολίες διότι δεν θα υπάρχει ο κατάλληλος αριθμός επαγγελματιών για να τροφοδοτήσουν το ίδιο τους το σύστημα. Ευχαριστώ, κυρία Χόιτοβα. Ευχαριστώ. Ε, χαιρετίζω αυτή την συζήτηση και ιδίω τη μελέτη διότι η μελέτη αυτή κατά τη γνώμη μου αποκαλύπτει ένα πολύ βασικό θέμα το οποίο μας απασχολεί όλους σε αυτή την αίθουσα και πρόκειται για την ε, σωστή χρονική στιγμή της εφαρμογής μιας οδηγίας. Ένα δεν καταλαβαίνω. Όλα τα, με, ε, όλοι τα κράτη-μέλη είχαν συμφωνήσει με την προθεσμία εφαρμογής και κανένα κράτος τελικά δεν σεβάστηκε την εφαρμογή. Οπότε τα κράτη-μέλη δεν ε, ε, εξετίμησαν σωστά τις δυνατότητές τους. Αυτό ήταν το πρώτο συμπέρασμα στο οποίο κατέληξα. Δεύτερον, η αιτία γι' αυτό κατ' εμέ είναι η εξής. Εν, ε, αντιθέσει με άλλες περιπτώσεις όπου είμαστε υποχρεωμένοι να ε, εφαρμόσουμε μια ολόκληρη σειρά οδηγιών και αποφάσεων στον τομέα της εκπαίδευσης ε, δεν υπάρχει συνήθεια να εφαρμόζονται οι οδηγίες. Ε, είναι ένας τομέας ο οποίος ρυθμίζεται συνήθως σε εθνικό επίπεδο, δηλαδή δεν υπάρχουν επαρκείς εμπειρίες με την εφαρμογή των ευρωπαϊκών οδηγιών και κατ' εμέ εκεί οφείλεται το πρόβλημα. Θα ήταν λοιπόν καλό και ε, να μπορέσουμε να πιέσουμε τα κρατη μερη να αλλάξουν συνήθειες και να συνηθίσουν και στον τομέα αυτό να εφαρμόζουν τις ε, οδηγίες εγκαίρως ε, όσον αφορά τις ικανότητες του υγειονομικού προσωπικού και δεν αναφέρομαι εδώ μόνο στους γιατρούς αλλά ιδίως στις νοσοκόμες και στους φυσιοθεραπευτές ε, πρέπει να υπάρχει μία ε, κινητικότητα στην εσωτερική αγορά και άρα πρέπει να πιεστούν τα κράτη-μέλη ε, διότι θα πρέπει να υπάρχει ένα συντονισμός για τις αποζημιώσεις του προσωπικού υγείας και δεν θα πρέπει το κίνητρο να είναι μόνο ο μισθός διότι οι μισθοί αποτελούν σε ένα θέμα της εσωτερικής αγοράς. Όλοι προσπαθούν να αγοράσουν φθηνότερα είτε δυνάμεις ε, ή εργατικό δυναμικό είτε προϊόντα. Ε, κάθε κράτος ρυθμίζει μόνο του τις μεθόδους τους και εγώ εμένα μου είπε ε, μία διευθύντρια νοσοκομείου ότι πολλές νοσοκόμες ζητούν εξηγήσει διότι υπάρχουν οι κανόνες ε, για την αναγνώριση των προσόντων και παρόλα αυτά έχουν ορισμένα διπλώματα τα οποία δεν καλύπτονται από, τα, ε, από την νομοθεσία και ε, υπάρχουν πάρα πολλά διπλώματα ιδίως για το, τις αδερφές και για το νοσοκομιακό προσωπικό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν είναι σαφής. Άρα δεν μπορούμε να εναρμονίσουμε την ε, την εκπαίδευση στον τομέα αυτό. Εάν είχαμε όμως μία τράπεζα δεδομένων και εκεί καταγράφαμε τα διάφορα διπλώματα θα μπορούσαν να βοηθηθούν και οι κρατικές αρχές και οι υπεύθυνοι στις άλλες χώρες ε, και να αξιολογήσουν αν η εκπαίδευση αυτή είναι ισότιμη ε, σε αυτές άλλων χωρών. Δηλαδή ε, η η νοσοκόμα χρειάζεται 30, 3 μήνες για να γνωρίσει αν θα αναγνωριστεί το δίπλωμά της και τι διαβήματα πρέπει να κάνει για να υπάρχει αναγνώριση του διπλώματό της. Νομίζω ότι κάτι πρέπει να γίνει διότι εδώ υπάρχει ακόμη μία μεγάλη έλλειψη. Κυρία Πρόεδρε, συμφωνώ πολλά από αυτά ελέγχθησαν, ιδίως με την κυρία Ρόιτοβα. Δεν παραγνωρίζω το περίπλοκο του θέματος λόγω της ευρείας προσέγγισης της οδηγίας, αλλά πρέπει να σας πω ότι κατά βάθος ενοχλήθηκα διαβάζοντας το κείμενο διότι το κείμενο αυτό δεν είμαι βέβαιος ότι κατάλαβα σωστά εάν η οδηγία μπορούσε να επιτύχει στην εφαρμογή της ή όχι. Νομίζω ότι ε, δεν, ε, δεν έχει επιτύχει λόγω των εμπειριών που έχουμε και των αντιδράσεων των επαγγελματιών στις χώρες μας οι οποίοι μας λέγουν ότι το σύστημα υγείας έχει αντιμετωπιστεί μεν γενικώ, αλλά το, η κατάσταση είναι ακόμη δύσκολη. Είναι δηλαδή ένα τυπικό παράδειγμα ένα κλασικό παράδειγμα για την κακή αντίληψη που έχουν ε, οι συμπολίτες μας για την Ευρώπη. Δηλαδή ένα θαυμάσιο πρόγραμμα, ε, μία ε, έξοχη οδηγία η οποία μπορεί να συμβάλλει στην Ευρώπη και στην ευρωπαϊκή ιδέα και συγχρόνως είναι τόσο περίπλοκη στην εφαρμογή της ώστε πρέπει κανείς να είναι πεπισμένος Ευρωπαίος για να πιστεί ότι η Ευρώπη προβαίνει σε μια διευκόλυνση της καθημερινής ζωής των Ευρωπαίων. Μεταξύ των προτάσεων και των παρατηρήσεων που διατυπώνονται μέσα στο έγγραφο για να απλοποιηθεί η κατάσταση, βλέπω ότι όλα οργανώνεται σε, ε, όλα σε τοπικό επίπεδο για να μην εφαρμοστεί η οδηγία. Δηλαδή ε, μετατίθεται αλλά δεν εφαρμόζεται διότι οι επαγγελματικές οργανώσεις ε, εκ της φύσεώς τους θέλουν να προασπιστούν τα κεκτημένα τους και δεν θέλουν να εξελιχθεί το επάγγελμά τους, δεν, ε, ε, δεν συμφωνούν τα λόμπις που, ε, στο να προχωρήσει η κατάσταση. Όλα δηλαδή αυτά αποτελούν βασικές τροχοπέδεις επιτόπου. Δεν ξέρω λοιπόν αν μία βελτίωση διοικητική δεν θα βελτίωνε την κατάσταση. Δηλαδή από τις λύσεις που θα ζητούσαμε να διαρευνήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήταν απλώς να διευκολύνει την ε, πρόσβαση για τον απλό Ευρωπαίο προς ένα σύστημα προσωπικής προσφυγής ε, εύκολης, ε, συγκεκριμένης, διότι βλέπω σε ιατρικό επίπεδο ότι αν οι γιατροί ή οι νοσοκόμες θέλουν να προασπίσουν τα δικαιώματά τους δεν ξέρουν τι να κάνουν. Και η Ευρώπη που έπρεπε να τους, να τους διευκολύνει εμφανίζεται σαν ένα τεράστιο βουνό που είναι το αντίθετο από αυτό το οποίο επιζητούμε. Μήπως λοιπόν, πρότασή μου είναι, θα μπορούσαμε στις επόμενες εβδομάδες, μήνες, χρόνια να ε, βρούμε ε, εύκολα εργαλεία τα οποία θα είναι προσβάσιμα για τον ε, πολίτη για να μπορέσει να προβεί σε ατομική προσφυγή, για να μπορέσει να εφαρμοστεί η οδηγία και το πνεύμα της. καλές ερωτήσεις, οι οποίες όντως πρέπει να απαντηθούν. Η κυρία Βάιλερ στη συνέχεια. Hm, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είδαμε και είδαμε στο, όταν ψηφίσαμε ότι θα ήταν πολλά τα προβλήματα αλλά πόσο μεγάλη δυστυπιστία θα υπήρχε δεν το είχαμε διαπιστώσει. Ευχαριστώ για τις διευκρινήσεις και έχω να κάνω τρεις ερωτήσεις. Η πρώτη είναι η εξής. Η μελέτη αυτή την οποία κάνατε θεωρείτε ότι είναι αντιπροσωπευτική όταν 3% των κρατών ε, δεν εμφανίζονται διότι δεν έχουν ακόμη εφαρμόσει τις διατάξεις. Πιστεύω ότι αυτό είναι πολύ προβληματικό διότι ε, όταν ε, ψηφίσαμε τρία κράτη ήταν ενάντια στην ε, οδηγία είχαν πει όμως ότι θα την εφαρμόζανε και συγκεκριμένα το Λουξεμβούργο όλα αυτά τα κράτη που είχαν τότε αμφιβολίες τώρα δεν την έχουν εφαρμόσει. Δεν ξέρω αν είναι πολιτική καθυστέρηση επειδή δεν τη θέλανε. Επίσης το σύστημα ήμι το οποίο δεν το γνώριζα. Ε, είναι γενικό ή είναι ένα δίκτυο μεταξύ κρατών. Θα μπορούσαν και πολίτες οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα αναγνωρίσεως διπλωμάτων να λάβουν από εκεί πληροφορίες για τους λόγους για τους οποίους το δίπλωμά τους δεν αναγνωρίζεται και το τρίτο θέμα σχετικά με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που αναφέρεται. Φαντάζομαι ότι ε, αυτές ε, ε, είναι ακόμη εκρεμείς ή υπάρχουν και άλλες. Δηλαδή υπάρχει υπερπροστατευτισμός, ανόητος υπερπροστατευτισμός, διότι βλέπουμε εδώ μηχανικούς, αρχιτέκτονες. Δεν φαντάζομαι ότι αυτοί δεν θα μπορούσαν να δουλέψουν σε άλλες χώρες. Πιο περίπλοκο είναι το θέμα για τα υγειονομικά επαγγελματικά επαγγέλματα διότι όπως είπε η κυρία Ρόιτοβα εις ε, το επαγγέλματα υγείας υπάρχουν περισσότερα προβλήματα εάν χώρες οι οποίες ε, ε, ήδη έχουν προβλήματα δεν ε, διευκολυνθούν για την παροχή υγειονομικών υπηρεσιών. Δηλαδή θα, δεν μπορούμε να εμποδίσουμε γιατροί να πάνε στην Ελβετία, στην Αγγλία, στη Σουηδία και κυρία Ρόιτοβ αυτό δεν έχει σχέση μόνο με το μισθό αλλά και με τις συνθήκες εργασίες, με την ιεραρχία αρχική πρόοδο, τη σταδιοδρομία και ε, για άλλα θέματα που επηρεάζουν ε, τους ε, επαγγελματίες υγείας που θέλουν να σταδιοδρομήσουν διότι στη Γερμανία, στη Σουηδία παραδείγματος χάρη πέρα του μισθού υπάρχει και το θέμα της προαγωγής και των συνθήκων εργασίας. Ίσως λοιπόν έχει προβλεφθεί να ξαναγίνει μία συζήτηση, ένα είδος ακρόασης για να δούμε από τη μία πλευρά πώς δεν θα περιορίσουμε την ελεύθερη διακίνηση και από την άλλη πώς θα εμποδίσουμε ε, και να δούμε τι κάνουν ορισμένα κράτη-μέλη για να ε, μην αποκλείουμε ορισμένες περιοχές και δεν αναφέρομαι μόνο στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία αλλά στη Γερμανία όπου ορισμένες περιοχές, σε ορισμένες περιοχές οι γιατροί δεν θέλουν να δουλέψουν και μόνο υποπίεση θα πάνε να δουλέψουν εκεί. Πώς θα ήταν δυνατόν λοιπόν στα πλαίσια της προβλεπόμενης ακρόασης να καλέσουμε και τους υπευθύνους του Συμβουλίου για θέματα παιδείας για να δούμε και επαγγελματικής κατάρτισης για να δούμε πώς μπορούμε να καταλύσουμε τα εμπόδια τα οποία υπάρχουν ακόμη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λέχνερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ και ε, την ε, ε, κυρία για την εξαιρετική έκθεση. Η κυρία Βάιλερ είπε ότι και εμείς στη συζήτηση αυτή είχαμε επεκταθεί πάρα πολύ. Το θέμα είναι πολύ δύσκολο διότι ο ίδιος πολίτης ο οποίος παραπονείται ότι δεν αναγνωρίζεται σε μία άλλη χώρα παραπονείται επειδή ήρθε κάποιος άλλος από κάποια άλλη χώρα χωρίς να έχει τα προσόντα. Υπάρχουν πάρα πολλές παραδόσεις και δομές στα κλάτη μελη και μπορούμε να δεχτούμε ότι χρειάζεται κάποιος χρόνος για να εφαρμοστούν όλα αυτά και νομικά και πρακτικά διότι και εμείς και η ίδια η οδηγία εξετάζει το θέμα της, ε, των αδικαιολογή των εμποδίων στον ανταγωνισμό ο πρέπει να λάβουμε υπόψη και την προστασία του καταναλωτή αλλά και αντιστρόφως η συζήτηση η οποία γίνεται και συμφωνώ με την κυρία Παβάνοβα ε, υπάρχει ένα πρόβλημα αλλά δυστυχώς ε, δεν είναι μόνο θέμα επαγγελματικών προσόντων και διπλωμάτων υπάρχουν και άλλες πτυχές ε, πολύ ενδιαφέρουσες αλλά διαφορετικές οι οποίες αναπτύσσονται εδώ. Ιδίω διότι δηλαδή οι εμπειρογνώμονε τα κράτη-μέλη δεν εμποδίζονται καθόλου από την ε, οδηγία να αλλάξουν τις διατάξεις σχετικά με τα προσόντα και να μειώσουν ή να αυξήσουν τον πύχη για τα προσόντα για ε, αναλόγως του αν χρειάζονται και πώς προσωπικό από άλλες χώρες. Βέβαια ένα είναι το δίκαιο και από την άλλη είναι η πρακτική, δηλαδή η πραγματικότητα και εμείς θα πρέπει στο μέλλον να απασχολήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με όλα αυτά τα θέματα. Έχω λοιπόν ερωτήσεις. Καταρχήν, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει κάτι να κάνει τώρα εναντίον των κρατών μελών που δεν έχουν μερικώς ή πλήρως εφαρμόσει τις διατάξεις αυτές και η κυρία Σιλβέστη είπατε ότι ορισμένα κράτη δεν έχουν ε, εφαρμόσει πλήρως. Τι εννοείτε ότι δεν έχουν καλυφθεί ορισμένοι τομείς ή είναι πιο σοβαρό και δεύτερον θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό ότι συνεχίζουν να υπάρχουν προσφυγές. Ιδίως πολίτες που πλήττονται προσφεύγουν και όλα αυτά θα έπρεπε να συγκεντρωθούν, να διαρθρωθούν και να καταλήξουν σε κριτήρια. Να δούμε αν είναι κάτι που μπορεί να γενικευθεί ή αν είναι ε, ε, αναγκαίο να υπάρξει μία τράπεζα δεδομένων με επισκοπήσεις και γενικές παρουσιάσεις και τι προσαρμογές χρειάζεται για να μπορέσει να εφαρμοστεί αυτή στην νομοθεσία. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω αγαπητοί συνάδελφοι ότι έχουμε 10 λεπτά μόνο στη διαθεσή μας ακόμα για το συγκεκριμένο θέμα της ημερησίας διάταξης. Και υπάρχει και η έκθεση της κυρίας Σάλτρ Μόζε που ακολουθεί. Γι' αυτό θα ήθελα να ζητήσω από τους συναδέλφους να είναι σύντομοι για να μπορέσουμε να ακούσουμε και την απάντηση της ε, Κομισιόν στο ερώτημα του κ. Γιουβέν για το άρθρο 51 της οδηγίας. Η κυρία Ράπτη έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι όταν κάνουμε τέτοιου είδους συζητήσεις, το πρώτο και κύριο είναι να είμαστε ειλικρινείς. Ε, θα προσπαθήσω να είμαι ειλικρινής, έστω και αν δεν ε, είναι ευχάριστα, τα όσα θα πω. Ε, το πρώτο έχει να κάνει με τη γλώσσα που χρησιμοποιούμε. Είναι μια γλώσσα την οποία είπε πολύ εύστοχα ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι μια γλώσσα που δεν την καταλαβαίνουν οι πολλοί πολίτες της Ευρώπης και θα πρέπει κάτι να κάνουμε γι' αυτό. Το δεύτερο είναι ε, το θέμα των επαγγελματιών και καταναλωτών. Κάθε ε, επαγγελματίας ο γιατρός, η νοσοκόμα, ο εκπαιδευτικός, την ίδια στιγμή προσφέρει υπηρεσία σε καταναλωτές. Άρα θα πρέπει να έχουμε και τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Με άλλα λόγια θεωρώ για παράδειγμα ότι τα νοσοκομεία δεν υπάρχουν για να εργάζονται οι γιατροί και οι νοσοκόμες. Τα νοσοκομεία υπάρχουν για να γίνονται καλά οι ασθενείς. Άρα οι γιατροί και οι νοσοκόμες τα προσόντα τους και όλα όσα προβλέπουμε θα πρέπει να λαμβάνουν πρώτα και κύρια υπόψη την εξυπηρέτηση του ασθενούς. Άρα θα πρέπει στο πλαίσιο της Ευρώπης οι ασθενείς σε όλα τα κράτη-μέλη να μπορούν να βρίσκουν την υγειά τους. Εάν για παράδειγμα πάρω το παράδειγμα που ανέφερε η συνάδελφος πριν από τη Βουλγαρία. Εάν ξαφνικά φύγουν οι μισές νοσοκόμες από τη Βουλγαρία, σημαίνει ότι οι Βούλγαροι ασθενείς έχουν ένα πρόβλημα. Πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Ένα παράδειγμα. Το θέμα της εκπαίδευσης. Ε, προέρχομαι από την Ελλάδα και είναι το κράτος που ακούσατε στην εισαγωγή ότι έχει κακές επιδόσεις. Ε, το θέμα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στην Ελλάδα μας απασχολεί πάρα πολύ. Και υπάρχει μια μεγάλη κουβέντα εκεί για το αν θα πρέπει να ενταχθεί στην υπόθεση της εσωτερικής αγοράς ή όχι. Και μέσα σε όλα αυτά και στους γιατρούς και στους μηχανικούς και στους αρχιτέκτονες και στους εκπαιδευτικούς, η κεντρική ιδέα είναι η απασχόληση. Ε, όλη η ιστορία βρίσκεται στην απασχόληση και στις δυνατότητες που υπάρχουν ή δεν υπάρχουν. Ε, από εκεί και πέρα ε, υπάρχει στο τέλος το θέμα των προσόντων. Νομίζω ότι κάποιες φορές τα προσόντα τίθενται γιατί πραγματικά πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχουν, αλλά κάποιες φορές από κάποια κράτη-μέλη, σε αυτά α, τολμώ να περιλάβω και το δικό μου, την Ελλάδα, τα προσόντα τίθενται με τέτοιο τρόπο ώστε να χρησιμοποιούνται ως φίλτρα που κλείνουν τη δυνατότητα για να έρθουν από το εξωτερικό άλλοι από τα άλλα κράτη-μέλη να εργαστούν. Και ολοκληρώνω κυρία Πρόεδρε ε, με το θέμα του άρθρου 15 της οδηγίας, το οποίο αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ένα από τα θέματα που είχα σημειώσει, που αφορά τη δημιουργία κοινών βάσεων επαγγελματικών προσόντων. Και θέλω να ρωτήσω εάν υπάρχει η, η γνώση, η πληροφορία σε σχέση με τις επαγγελματικές ενώσεις και το πόσο διατεθειμένες είναι να προχωρήσουν σε κοινέ βάσεις. Και ε, αναφέρω ένα παράδειγμα, το θέμα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ενώσεως Ψυχολόγων. Και βεβαίως κλείνω με το θέμα της Ευρωπαϊκής Επαγγελματική Κάρτας, που νομίζω ότι οι κοινέ βάσεις είναι προϋπόθεση για την Ευρωπαϊκή Επαγγελματική Κάρτα, που εάν καταφέρουμε να γίνει πραγματικότητα, ε, νομίζω ότι θα βοηθήσει. Ευχαριστώ. Thank you Κύριος Κέλλη και μετά Κορέα. Ευχαριστώ, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Πάντα θεωρούσα ότι αυτή η οδηγία και η εφαρμογή της θα ήταν δύσκολη. Είναι η ανθρώπινη φύση τέτοια ούτως ή άλλως. Ε, η κυρία Γουίλερ πίσω μου αναφέρθηκε στο στο στάδιο εφαρμογής ε, της οδηγίας στα διάφορα κράτη-μέλη. Το πρόβλημά μου είναι, είναι αλήθεια, είναι, πραγματικά όντως έχει εφαρμοστεί η οδηγία αυτή και σε αυτό το βαθμό ή απλώς είναι λόγια. Ε, οι προθεσμίες ούτως ή άλλως που, είχε, ε, που προέβλεπε η οδηγία ήταν ιδιαίτερα φιλόδοξες ε, και ιδίως στον τομέα των, της, ιατρικό και των υγειονομικών. Ήθελα να ξέρω ε, έχουν αυξηθεί πολύ οι δυσκολίες. Όλα τα κράτη-μέλη δεν εφάρμοσαν την, ε, την οδηγία εγκαίρως. Αυτό σημαίνει ότι ε, δεν υπάρχει σεβασμός στις, ε, στις προθεσμίες και δεν υπάρχει σεβασμός στα όσα αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένω, είναι θέμα ε, συνολικό πιστεύω και συνολικής εμπιστοσύνης προς, προς τα όσα πρεσβεύουν και επιβάλλουν οι, οι, οι ευρωπαϊκές κοινότητες. Εδώ πιστεύω ότι υπάρχει ένα θέμα εμπιστοσύνης. Υπάρχουν κάποια στεγανά και θα πάρει πάρα πολύ χρόνο για να καταργηθούν αυτά και να ξεπεράσουμε τις καχυποψίε του παρελθόντος. Τώρα, Υπάρχει ένα βασικό σημείο το οποίο θα πρέπει να... Μάλλον πιστεύω ότι αυτή η οδηγία είναι πάρα πολύ σημαντική. Πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα. Το πρόβλημα είναι και η χρήση της γλώσσας. Χρειάζεται μια απλή γλώσσα για να μπορέσουμε να ε, εφαρμόσουμε κάποια κείμενα στην Ευρώπη και πιο συγκεκριμένα και αυτό το κείμενο που έχουμε μπροστά μας. Διότι αυτή η, η ευρωπαϊκή γλώσσα, αν θέλετε, η κοινοτική γλώσσα που χρησιμοποιείται, δυσκολεύει την κατάσταση. Τώρα, το σύστημα το, το οποίο χρησιμοποιείται για την, για την εσωτερική αγορά Ε, είναι ένα σύστημα μένα. όμως δυστυχώς δεν μπορέσαμε να το εφαρμόσουμε ποτέ έτσι όπως θα έπρεπε και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Ο κύριος Γιούβεν είπε ότι χρειαζόμαστε μια απλή διαδικασία για τους πολίτες οι οποίοι πραγματικά θλίβονται και ε, ε, έχουν, αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω της μη σωστή εφαρμογής της οδηγίας αυτής. Αυτό πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει. I think we all collective... Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές όμως. Εκεί καταλήγω. Διότι οι προθεσμίες που είχαμε υιοθετήσει δεν ήταν ρεαλιστικές. Και δείτε που μας οδήγησαν ο κύριος Κορέα. Είδαμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Άρα η συζήτηση αυτή και η έκθεση αυτή που μας παρουσιάστηκε τώρα ε, μας βοήθησε, γιατί συνειδητοποίησαμε την ύπαρξη του προβλήματος. Μετά, Πιστεύω ότι δεν έχουμε αρκετά εργαλεία στη διάθεσή μας ε, για να μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί. Επίσης, θα θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε και να εφαρμόσουμε την ελεύθερη κυκλοφορία ανθρώπων και αγαθών. Η ελεύθερη κυκλοφορία είναι ένα βασικό στοιχείο για την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς. Θα πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη μας και το ανθρώπινο δυναμικό, τους ανθρώπινους πόρους. πρέπει, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τι δεν πήγε στραβά για να το διορθώσουμε. Και απευθύνομαι τώρα στην Κομισιό. Η Κομισιό εξετάζει το όλο θέμα μέσα στα πλαίσια της ελευθερίας ε, διακίνησης. Όμως δεν το βλέπουν από την πλευρά της αγοράς. Εγώ πιστεύω ότι ανεξάρτητα από προβλήματα επικουρικότητας θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ναι μεν υπάρχει προσφορά και ζήτηση σε εθνικό επίπεδο, άρα το θέμα της επικουρκότητας είναι σημαντικό, αλλά θα πρέπει να μπορούμε να συγκρίνουμε τις πληροφορίες που αφορούν και την στρατηγική οργάνωση των ανθρωπίνων, δικαιωμάτων, των ανθρωπίνων πόρων σε κάθε χώρα. Ε, θα πρέπει να γίνει μια τράπεζα δεδομένων ενδεχόμενα. Ε, θα Πρέπει να έχουμε συγκεκριμένες και μονοποιημένε πληροφορίε για το τι ισχύει για κάθε επάγγελμα σε κάθε χώρα. Ευχαριστώ. Η κυρία Ρούλε, θα είσαστε σύντομοι φαντάζομαι. ένα θέμα το οποίο δεν έχει αναφερθεί και θα ήθελα να επανέλθω σχετικά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατέκρινε το θέμα του Single Contact Points. Προτού λοιπόν προτείνει Single Contact Points στο, σε μελλοντική οδηγία, θα ήταν καλό να κοιτάξει τις ε, διαρθρωτικές δομές στα κράτη-μέλη για να δει μήπως ε, η διοικητική δομή των κρατών καθιστά το θέμα πολύ περίπλοκο γιατί με ενόχλησε αυτό που είπε. Επίσης Νομίζω ότι ένα, ε, μια δημόσια τράπεζα δεδομένων θα μπορούσε να βοηθήσει διότι σε ορισμένα κράτη υπήρξε πίεση προς ε, τους ενδιαφερομένους ε, από όταν άρχισε να συζητείται η αμοιβαία αναγνώριση διπλωμάτων. Πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα που να είναι διαφανές, διότι πρόκειται ε, για καταχρήσεις. Δεν, δεν είναι φυσιολογικές πρακτικές και θα έπρεπε κανείς να τις αποδυναμώσει. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα, ετέθησαν πάρα πολύ καλές ερωτήσεις. Ε, τα θέματα που αφορούν ε, στο άρθρο 15, στο άρθρο 51. Να δώσω λοιπόν ε, το λόγο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην κυρία Σίλβες. Καταρχάς, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κυρία Πρόεδρε, επειδή είναι περιορισμένος ο χρόνος, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Το πρώτο θέμα το οποίο θα ήθελα να θίξω είναι ότι έγιναν πολλές ερωτήσεις για το εάν η οδηγία αυτή είναι αποτελεσματική και βοηθά τον πολίτη. Ουσιαστικά εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει για όλες τις οδηγίες που προβλέπει και είναι κάτι που θα ξεκινήσουμε υπό την ε, νέα Επιτροπή. Αν, αν ε, ε, άκουσα σωστά τον κύριο Μπαρόζο την περασμένη εβδομάδα θα γίνεται ex post αξιολόγηση, εκ των υστέρων αξιολόγηση δηλαδή. Βλέπετε λοιπόν εγώ είμαι προσεκτικός σε αυτά που λέω, εσείς θα πρέπει να ε, προβείτε στις ερωτήσεις για να κινητοποιηθούμε. Αναφερθήκατε στην κινητικότητα του προσωπικού σε όλο τον τομέα, ιδίως όσον αφορά τους γιατρούς και τις νοσοκόμες είναι προφανές ότι έχουμε ένα κεκτημένο σχετικά με αυτόν τον ε, ε, ιατρικό χώρο που εναρμονίζει ε, το πεδίο. Υπάρχει και το οποίο όμως υπάρχει εδώ και 30 χρόνια. Και ποτέ δεν σκεφτήκαμε εάν θα έπρεπε να αξιολογηθεί, αν θα έπρεπε να αναθεωρηθεί. Αυτή τη στιγμή παρακολουθούμε προσεκτικά τη συζητήσεις για τη συνθήκη της Λισοβόνας, γιατί αν ισχύσει ε, προβλέπεται ότι χρειάζεται ομοφωνία με αυξημένη πλειοψηφία στο Συμβούλιο. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί είμαι πολύ προσεκτικός για το πώς μιλάω. Ε, για τα δύο χρόνια θα έπρεπε σε αντίθεση με την ε, οδηγία παροχής υπηρεσιών ε, να πούμε ότι 80 ή 90% υπήρχε ήδη στο κεκτημένο προτού ισχύσει αυτή η οδηγία. Εάν το συγκρίνουμε ιδίως με την οδηγία παροχής υπηρεσιών, ε, εδώ πολλά προϋπήρχαν. Το άλλο θέμα το οποίο θα ήθελα να αναφέρω είναι τα δικαιώματα των πολιτών και μιλάμε για το ατομικό, την ατομική προσφυγή στο άρθρο 51 ε, και την τράπεζα δεδομένων. Σήμερα δεν μπορώ να σας πω ακριβώς πώς λειτουργεί ακριβώς το άρθρο 51 η διάταξη υπάρχει, ε, κοιτάμε τα κράτη-μέλη να την εφαρμόσουν και οι ε, πολίτες να γνωρίζουν τι δικαιώματα έχουν για να προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Εάν υπάρχει ένα σύστημα πληροφοριών, όχι διότι πολλά ελέγχθησαν ε, περί μίας τράπεζας δεδομένων η οποία υπάρχει, υπάρχει στην ιστοσελίδα μας και έχει ήδη πολλά στοιχεία. Αναφερθήκατε επίσης στο θέμα των σημείων επαφής. Συμφωνώ. Δεν θέλω να κατακρίνω τις ε, επαφές, αλλά εάν ε, μιλούμε στην οδηγία για κάτι, πρέπει να γνωρίζουμε ότι θα λειτουργεί σε εθνικό επίπεδο και σε δημοσιονομικό επίπεδο. Γι' αυτό και αυτή τη στιγμή η ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ευχαρίστως είναι στη διάθεσή σας αλλά θα πρέπει ο πολίτης να διευκολυνθεί να μην χρειάζεται να αναλάβει το μακρύ δρόμο στη δικαιοσύνη και επίσης ε, είπατε τι κάνουν τα κράτη-μέλη για να προωθήσουν τα θέματα αυτά και αν εφαρμόζουν το, τις διατάξεις. Ελπίζομαι το Νοέμβριο να δείξουμε έναν πίνακα βαθμολογίας, ε, ένα scoreboard. Ξέρετε το internal market scoreboard, αλλά εμείς το Νοέμβριο σκοπεύουμε να κάνουμε έναν πίνακα βαθμολογίας όπου θα δείξουμε πού βρίσκονται τα κράτη πότε θα πρέπει να γίνει η τελική εφαρμογή διαφόρων διατάξεων. Παραδείγματο χάρη το ίδιο ε, θα ισχύσει και για την οδηγία παροχής υπηρεσιών. Τι γίνεται με τους ε, ψυχολόγους. Το ερώτημα ήταν αν είναι ρυθμισμένο το επάγγελμα των ψυχολόγων στα κράτη-μέλη και χρειάζεται ένα σημείο εκκινήσεως για την ελεύθερη διακίνηση. Πρέπει κανείς να βοηθήσει και ε, να κοιτάξει να βελτιώσει ότι υπάρχει σε κάθε κράτος. Την άλλη εβδομάδα θα δω τους ψυχολόγους και θα κάνω ε, μία συζήτηση. Μιλήσαμε για ακρόαση, αλλά αυτή εξαρτάται από το τι θέλει να κάνει το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ για την προσοχή σας και δεν θέλω τώρα να καταχρεστώ το χρόνο σας. Ευχαριστώ, κυρία Σίλβιτ. Ευχαριστώ και εγώ θα είμαι πολύ σύντομη και θα απαντήσω απλώς σε ερωτήσεις που απευθύνθηκαν σε μένα. Η κυρία Βάιλερ είχε κάποιες ερωτήσεις. Κατά πόσον είναι αντιπροσωπευτική αυτή η μελέτη, θα μπορούσα να πω ότι ναι, μιλήσαμε με εθνικά σημεία επαφή και εθνικού συντονιστέ σε όλα τα κράτη-μέλη. Επομένω, όντω καλύπτει τα πάντα και έχουμε πληροφορίες από όλα τα κράτη-μέλη. Για το IMI, το σύστημα αυτό, το οποίο αναφέρθηκε ήδη και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το κατά πόσον υπάρχει πρόσβαση για τους πολίτες. Δεν νομίζω ότι σκοπό έχει τους πολίτες. Είναι ένα σύστημα για να βοηθήσει τους επαγγελματίες. Ε, αυτό που έχουν οι πολίτες είναι το δίκτυο Solvent που έχει πολλές εθνικές πληροφορίες και ε, παρέχει συνδρομή απευθείας στους πολίτες. Έχουν πολύ καλό σημείο εισόδου, αν θέλετε, εκεί. Επίσης αναφερθήκατε και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ε, το κατά πόσον έχουμε όλες τι αποφάσεις ή περιμένουμε και άλλες. Οι υποθέσεις που μπορεί να ασχοληθεί το δικαστήριο και αφορούν και την Επιτροπή σας εδώ είναι ε, καθυστερήσεις ή τα μέτρα τα οποία λήφθησαν για την ε, μεταφορά της οδηγίας. Πολλές από αυτές οι υποθέσεις εκκρεμούν. Τώρα, προσφυγές ε, για μεμονωμένα άτομα σαφώς θα προκύπτουν συνεχών, συνεχώς, αλλά δεν τις έχουμε λάβει υπόψη σε αυτή τη μελέτη. Έχουμε, τις έχουμε λάβει υπόψη, αλλά δεν ε, υπάρχουν ε, προσφυγές με τις οποίες ασχοληθήκαμε. Η κυρία Ράπτη ρώτησε κατά πόσον έχουμε περισσότερο πληροφορίες για τους συνδέσμους επαγγελματιών και κάποια κοινή βάση ή κάποιο κοινό πιστοποιητικό. Υπάρχουν κάποια παραδείγματα, αναφερθήκατε και στους ψυχολόγους, οι οποίοι είναι όντως ε, υπέρ κάποιου ενιαίου ευρωπαϊκού πιστοποιητικού για τους ψυχολόγους και προτείνεται όντως ε, κάτι αντίστοιχο, ε, κάποιες επαγγελματικές κάρτες. Δεν μπορώ να σας πω κάτι για το κατά πόσο αυτή είναι η τρέχουσα τάση μεταξύ των επαγγελματικών ομάδων, αλλά νομίζω ότι αρκετού τι από αυτούς είναι υπέρ Τη δημιουργία ε, κάποιου στοιχείου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά έχουμε μιλήσει με ελάχιστου. επομένως δεν μπορώ να σας πω κάτι συγκεκριμένο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση. Γιατροί, νοσοκόμες, ε, είναι αυτοί στους οποίους σταθήκαμε. Ως ακαδημαϊκή φιλόσοφος ε, διαπίστωσα ότι δεν αναφέρθηκε κανένας φιλόσοφος. Ποια θα ήταν η αμοιβαία αναγνώριση μεταξύ ενός ε, Φιλανδού και Έλληνα φιλοσόφου. Τέλος πάντων, ευχαριστώ πολύ τους εμπειρογνώμονες και τους καλούς συναδέλφους για τις ε, πολύ καλές τους ερωτήσεις. Το επόμενο θέμα πολύ ενδιαφέρον και πολύ νόστιμο. Αφορά πληροφορίες ε, για τρόφιμα στους καταναλωτές. Είναι ακριβώς πριν από το γεύμα. Να δώσουμε το λόγο στην κυρία Σαλδεμόζε, αλλά νομίζω ότι κάτι ήθελε να μας πει η γραμματεία. Όχι. Ωραία. Κυρία Σαλδεμόζε, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Την τελευταία φορά που συζητήσαμε, που συναντηθήκαμε. Συζητήσαμε το θέμα αυτό και κυρίως μέσα στα πλαίσια της προηγούμενης θητείας και μέσα στα πλαίσια μιας α, κοινή έκθεσης είχαμε ψηφίσει κιόλας για το θέμα αυτό. Να περιμένω λίγο να καθίσουν όλοι, να τακτοποιηθούν και μετά να συνεχίσω. Quickly move. We will let Mrs. to speak. Øh, Ωραία, συνεχίζω. Λοιπόν, έχουμε ψηφίσει μία γνωμοδότηση μαζί με την Επιτροπή Περιβάλλοντος που είναι η επί της ουσίας αρμόδια επιτροπή. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος όμως αποφάσισε να ξεκινήσει ξανά και να ζητήσει γνωμοδοτήσει ε, ξανά από, από μια ολόκληρη σειρά επιτροπών. Γι' αυτό το λόγο μας δίδεται αυτή η ευκαιρία και σε εμά να συζητήσουμε για τα θέματα που αφορούν τα τρόφιμα. Και μετά έχουμε και τα νέα μέλη που θα θέλανε ε, προφανώς να μας πούνε τις απόψεις τους. Όμως ας δούμε ποιο είναι το, ποια είναι το, πιο το χρονοδιάγραμμα στην Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, θα σας πω ότι εμείς εγώ τι προτίθεμαι να κάνω και θα δούμε μετά. Να συζητήσουμε και το περιεχόμενο της έκθεσής μας και να δούμε πού θα πάμε από εδώ και πέρα. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος έχει ορίσει την Ρενάτα Σόμερ σαν εισηγήτρια και για άλλη μια φορά και αυτή έχει κάνει κάποιες προτάσεις σύμφωνα με τις οποίες η Επιτροπή Περιβάλλοντος θα υιοθετήσει την έκθεση της τον Μάρτιο του 2010. Και φαίνεται ότι θα ψηφίσουμε τον Μάιο του 2010. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα το οποίο έχουμε, το οποίο πρέπει να ακολουθήσουμε. Αυτό το οποίο προτείνω επομένως είναι να συζητήσουμε σωστά και ήρεμα την ε, επιτροπή, στην Επιτροπή μας το θέμα αυτό. Πρώτη Δεκεμβρίου μπορούμε να συζητήσουμε την έκθεσή μου, διότι 11 Νοεμβρίου θα τη στείλω για μετάφραση. Επομένως θα έχουμε μια προθεσμία υποβολής τροπολογιών μέχρι 6 Ιανουαρίου, ε, θα τη συζητήσουμε μέχρι τις 25 Ιανουαρίου και μετά στις 23 Φεβρουαρίου να ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας την έκθεση. Έχουμε, θεωρώ, αρκετό χρόνο με τον τρόπο αυτό στη διάθεσή μας για να συζητήσουμε το θέμα. Όλα αυτά όμως εξαρτώνται ε, από, το, από μια προϋπόθεση, δηλαδή ότι υπάρχουν τροπολογίες, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρόκειται για μια έκθεση η οποία ήδη υπάρχει, η οποία, για την οποία, την ε, άρα μπορούμε να επιταχύνουμε κάπως ε, τα πράγματα, γιατί θα πρέπει να δούμε και με τους άλλους συνεισηγητές ε, τι χρειάζεται να αλλάξει από την γνωμοδότηση αυτή. Τώρα, ποιο είναι το θέμα μας έκανε η Κομισιόμια μια πρόταση για, την, για τις πληροφορίες που αφορούν τα τρόφιμα και η πρόταση αυτή έχει σαν στόχο να συγκεντρώσουμε όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται στα διάφορα νομοθετικά κείμενα για την ετικετοθεσία, για την ασφάλεια τροφίμων κτλ. Και όλα αυτά συμπεριλαμβάνονται σε αυτό, σε αυτό το κείμενο. Δύο στοιχεία βασικά υπάρχουν εδώ. Το ένα είναι η ετικετοθεσία, η σχετική επισήμανση των ε, τροφίμων. Τι πληροφορίες πρέπει να αναφέρονται πάνω στην, ε, στη συσκευασία, ε, για αλλεργιογόνα, για χώρες προέλευσης κτλ. κτλ. Αυτά αφορούν το γενικό κομμάτι. Και μετά θα πρέπει να Υπάρχουν πληροφορίες για τα ε, διατροφικά στοιχεία, δηλαδή ε, στοιχεία τα οποία πρέπει να είναι οπωσδήποτε πάνω στην ε, συσκευασία. Για τις θερμίδες, για την περιεκτικότητα σε διάφορα λιπαρά, πρωτεΐνες κτλ. Όλα αυτά τα διατροφικά στοιχεία πρέπει και οι πληροφορίες πρέπει να αναφέρονται ε, στην, ε, στη συσκευασία. Υποχρεωτικά. Υποχρεωτικά τονίζω. Τώρα, στην αρχική γνωμοδότηση είχαν υποβληθεί, είχαν υποβληθεί ένας τεράστιος αριθμός πληροφοριών και πραγματικά ε, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να καταλήξουμε σε μια κοινή θέση με βάση τις τροπολογίες που είχαν υποβληθεί. Τα καταφέραμε βέβαια γιατί τελικά μπορέσαμε να συνοψίσουμε όλες αυτές τις τροπολογίες σε 10 συμβαστικές τροπολογίες. Υπήρξε συμφωνία, παραδείγματο χάρη, στα θέματα και τα διατροφικά, όταν μιλάγαμε για το περιεχόμενο να μιλάμε σε, σε 100, με βάση 100 γραμμάρια 100 μιλιλίτρια και όχι με βάση το ένα, κάποιο ποσοστό. Επίσης είχαμε συμφωνήσει ότι θα έπρεπε να διευρύνουμε τον κατάλογο των ε, συστατικών που θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνονται και μετά υπήρξε και μια συμβιβαστική, και μια συμβιβαστική πρόταση για άλλα υποχρεωτικά στοιχεία, για άλλες υποχρεωτικές πληροφορίες παραδείγματος χάρη η, η ημερομηνία παραγωγής, εάν υπήρξε κάποια ε, επεξεργασία στην επιφάνεια, εάν πρόκειται για φρούτα παραδείγματο χάρη. Επομένως η δουλειά ήταν πάρα πολύ σημαντική ε, που είχε γίνει σε επίπεδο επιτροπής και υπήρξαν πραγματικά αρκετές συμβαστικές τροπολογίες που αντικατόπτριζαν ε, τις απόψεις όλων. Τώρα, η καινούργια γνωμοδότηση θεωρώ, η καινούργια έκθεση θεωρώ δεν, έχει μεγάλες διαφορές σε σχέση με την προηγούμενη. Εξαρτάται βέβαια όμως από την Επιτροπή αυτό. Υπάρχουν κάποιες αλλαγές που θα ήθελα βέβαια και εγώ να γίνουν. Ε. Το GDA, ε, Guideline Daily Amounts, η, η, η, ε, τα οι, οι ποσότητες, οι ημερήσιες μερίδες, τέλος πάντων, οι προτινόμενες, ε, οι προτινόμενες ημερήσιες μερίδες. Διο... Διορωτώ με πως έπρεπε να το βγάλουμε αυτό απ' έξω. Αυτό τον εθελοντικό χαρακτήρα, να τον, τον προαιρετικό χαρακτήρα να τον αφαιρέσουμε. Και έγινε μια μεγάλη κουβέντα για το κατά πόσον το να αναφέρουμε πάνω σε μια συσκευασία το ποσοστό της προτινόμενης ημερήσιας ε, μερίδας ε, βοηθάει το καταναλωτή ή όχι. Γιατί οδηγούμεθα σε κάποια παράδοξα. Δηλαδή ότι ας πούμε ένα πράσινο μήλο είναι λιγότερο θρεπτικό από ότι μια, μια, ένα, μια, μια ποσότητα ας πούμε cornflakes που έχουν και ζάχαρη κιόλας. Γι' αυτό θα πρέπει να το, να το δούμε αυτό ίσως από κάποια διαφορετική σκοπιά για τις ημερήσιες προσλαμβανόμενες ε, ποσότητες. Τέλος πάντων, θα πρέπει να δούμε επίσης ε, και την άποψη των σκιωδών ε, εισηγητών, να δούμε δηλαδή κατά πόσον ε, θα πρέπει να αλλάξουμε ριζικά τη γνωμοδότηση ε, ή θα πρέπει να παραμείνουμε στην, σε ένα μεγάλο βαθμό σε αυτά που ήδη έχει, έχει καταλήξει η προηγούμενη εισηγήτρια. Τώρα, επίσης θα ήθελα να ξέρω, το χρονοδιάγραμμα που σας πρότεινα σας ικανοποιεί, μας αφήνει αρκετό χρόνο. Αυτά είχα να πω επί του παρόντος. Ε, είμαι στην διάθεση όλων των συναδέλφων ε, γιατί θα ήθελα πραγματικά να συνεργαστούμε όλοι μαζί. Και θα ήθελα τώρα να ακούσω και τις απόψεις σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και εδώ σε αυτήν την οδηγία θα πρέπει να τονίσουμε ορισμένες αρχές. Για τον καταναλωτή πρέπει να δίδονται πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να είναι σαφείς, ε, κατανοητές, αναγνώσιμες και θα πρέπει το κόστος της πληροφορίας να μην οδηγήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις εκτός αγοράς διότι οι πληροφορίες οι οποίες πρέπει να δώσουν οδηγούν στο ότι συνεπάγονται τεράστιες δαπάνες. Γενικώ η εργασία αυτή είναι σωστή. Οι ε, καταναλωτές πρέπει να πληροφορούνται χωρίς να κατακλείζονται. Ε, αυτά λοιπόν τα οποία ε, τους δίνουμε τώρα είναι κάπως υπερβολικά. Αν μπορούν να γνωρίζουν ποιες είναι οι θερμίδες, τι σχέση έχει με την ε, καθημερινή θρεπτική ουσία, τι είναι το ποσοστό άλατος ε, και πώς συνδυάζεται με την ε, ημερήσια πρόσληψη άλατος είναι βασικές πληροφορίες. Θα πρέπει λοιπόν αυτή η οδηγία να περιέχει και ορισμένους ορισμούς κατά τρόπον ώστε ο ο παραγωγός να μην μπορεί να εμφανίζει ό,τι θέλει πάνω σε μια τέτοια πινακίδα. Θα πρέπει η οδηγία ε, να καθορίζει τη βάση επί της οποίας θα πρέπει να προσφέρονται οι πληροφορίες. Εάν η πληροφόρηση είναι σαφής και ως το δυνατόν λιγότερο δαπανηρή, τότε θα έχουμε πετύχει. Είναι πολύ βασικό ε, να κάνουμε ένα βήμα για να ε, ε, καταστήσουμε την εσωτερική αγορά ενιαία, διότι πολλές επιχειρήσεις απευθύνονται στην εσωτερική αγορά και θα πρέπει να μπορούν να προσφέρουν τα προϊόντα τους ενιαία σε ολόκληρη την ενιαία αγορά και γι' αυτό θα πρέπει να έχουν συνεκτικά στοιχεία. Ευχαριστώ. Η κυρία Ρόλε. Ήμουν σκιώδης την προηγούμενη φορά και εγώ ξέρω ότι αυτά τα, αυτές οι 280 τροπολογίες με είχαν επιβαρύνει. Ε, ε, ε, ήταν πολύ τεταμένη η κατάσταση οπότε εγώ θα έλεγα να θεωρήσουμε σε βάση την έκθεση Ντανιό, να δούμε δηλαδή ε, πού έχουμε προβλήματα με την έκθεση Ντανιό και τι μπορούμε να διατηρήσουμε από την προηγούμενη έκθεση. Δεν είναι δηλαδή αναγκαίο να ξεκινήσουμε πάλι από την αρχή. Υπάρχουν ε, συμβιβαστικές λύσεις οι οποίες δεν θα διαφέρουν τόσο πολύ από τις προηγούμενες και θα χάσουμε χρόνο. Όσον αφορά τα GDA, ε, πιστεύω ότι θα πρέπει να τα συσχετίσουμε με προϊόντα που είναι αποτέλεσμα επεξεργασίας. Εκεί έχουμε το πρόβλημα στα μεταποιημένα προϊόντα και όχι παραδείγματο χάρη στις πατάτες. Ευχαριστώ κύριε Σουάμπ, θέλετε να μιλήσετε σας και όχι, η κυρία Κέρμερ τότε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θεωρώ ότι το θέμα των τροφίμων είναι πολύ ενδιαφέρον και εγώ θα ήθελα να το ξανασυζητήσουμε, διότι υπάρχουν και νέοι συνάδελφοι και γι' αυτό θεωρώ ότι δεν είχα διαβάσει με αρκετές λεπτομέρειες την πρώτη φορά την έκθεση και θα πρέπει σε ορισμένα θέματα να τα αναθεωρήσουμε. Σας λέω όμως ποιες είναι οι βασικές μου ιδέες, διότι είναι ένα θέμα στο οποίο συμφωνούμε όλοι. Δηλαδή υπάρχουν και συγκεκριμένες διατυπώσεις που έχω να προτείνω όσον αφορά ε, τον χαρακτηρισμό των τροφίμων και είναι θέματα που μπορούμε να περιλάβουμε εδώ και θα αποτελέσει ένα, μία ένδειξη διότι ε, θα υπάρχει μία σαφής ε, ρύθμιση και θα χαιρόμαστε. Ήμουνα ιδιαιτέρως αν μπορούμε να συνεργαστούμε μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Ένα θέμα που μας ενδιαφέρει όμως ίσως πιο πολύ και εδώ θα ήθελα να αναφερθώ εις τον εκπρόσωπο των φιλελευθέρων θα πρέπει ε, να λάβουμε υπόψη αυτό που είπε και η κυρία Ρούλε δηλαδή όσον αφορά τα επεξεργασμένα προϊόντα και όχι τις φυσικές ουσίες ε, ε, όσον αφορά τα θέματα αυτά πρέπει να σας πω ότι εγώ για τα GDA σύμφωνο διότι πιστεύω ότι όταν κοιτάζω ένα προϊόν, μία πίτσα παραδείγματο χάρη, με την πρώτη ματιά μπορώ να διαβάσω τι ποσοστό έχει ζάχαρη, αλατιού, και ε, αν έφαγα το μεσημέρι μίας, ε, μία πίτσα, αν ξέρω και τις θερμίδες, αφού το βράδυ μία, θα, ε, μία σαλάτα. Εάν όμως έρχει ένα πακέτο και πρέπει σε κάθε ταμπλέτα να υπάρχουν όλες οι λεπτομερές ενδείξεις, μπορεί κάποιος να μου πει για ένα προϊόν προϊόν το οποίο δεν είναι ε, ίσως τόσο ακριβώς περιγεγραμμένο ότι α, α, είμαι κάτω από το όριο, μπορώ να φάω 3, 4, 5 κομμάτια και ε, να έχω ξεπεράσει το όριο. Θα έπρεπε λοιπόν καλύτερα να ξέρουμε ποιες είναι οι ημερήσιες τιμές τις οποίες μπορεί να καταναλώσει κανείς. Υπάρχουν ορισμένοι στο Κοινοβούλιο οι οποίοι λένε ας έχουμε μόνο ε, στην πρώτη σελίδα τις θερμίδες και μόνο τα απόλυτα στοιχεία όπως η κυρία Ζόμερ παραδείγματο χάρη. Αλλά εγώ πιστεύω ότι τα GDA είναι καλά μέση τοποθέτηση είναι και η θέση της Υπουργού μας κατανάλωσης και εγώ πιστεύω ότι αυτή η μέση ε, κατάσταση είναι καλύτερη. Ε, όπως ε, παραδείγματο χάρη το παράδειγμα για το μήλο και το μουσλι εγώ δεν το κατάλαβα διότι μπορώ πάνω στην ετικέτα να δω και για το μουσλι πόσο χρειάζομαι σε ποσοστό της, ενιαία, της μου κατανάλωσης ενώ το μήλο δεν χρειάζεται να το καταγράψουμε διότι είναι ένα φυσικό προϊόν. Δεν κατάλαβα σε τι αποσκοπούσε το σχολείο σας αυτό. Ε, θα τραβούσα τη γραμμή ε, όσον αφορά τα προσθετικά και τις, προσε... Ε, τις ουσίες που προστίθενται διότι κατά τα άλλα συμφωνώ απολύτως με το να προωθήσουμε τα GDA. Mr. Ταραμπέλα, please. Ο κύριος Ταραμπέλα. Bien, je crois qu'en cette matière particulièrement sensible. Νομίζω ότι για αυτό το θέμα που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο, θα πρέπει να αποφύγουμε αυτό το ότι το, καλό είναι εχθρό του ε, καλύτερου. Μάλλον το καλύτερο είναι εχθρό του καλού. Ε, θα πρέπει να χρησιμοποιούμε καταρχάς μια, ένα μια ενιαία ποσότητα αναφοράς, 100 γραμμάρια, 100 μιλιλίτρια κτλ. Και εκεί να λέμε αυτή είναι η περιεκτικότητα ζάχαρη κτλ. Τώρα από εκεί και πέρα, να, βάζ, να λέμε εντάξει, είναι, έχει πολύ ζάχαρη, έχει λιγότερη ζάχαρη, δεν έχει καθόλου ζάχαρη, είναι ένα πράγμα. Αλλά σε σχέση με την προτινόμενη μερίσια πρόσληψη, να σας πω ότι είμαι ε, πολύ διστακτικός. Εξαρτάται από το άτομο. Εγώ, ας πούμε, ε, όταν βλέπω τα chips πρέπει να, να, να, τρέχω μακριά. Είναι 700, 700 ερμίδες 100 γραμμάρια. Αλλά βλέπω ότι υπάρχουν γύρω, γύρω, γύρω μου άτομα τα οποία ε, και λίγες παραπάνω σελίδες να καταναλώσουν δεν θα, δεν, θα τους βλάψουν. Δηλαδή εξαρτάται από το, από το πώς είναι ο καθένας. Από την άλλη πλευρά και αν έχει κάποια ασθένεια, Α πούμε, ο διαβητικός θα πρέπει να προσέχει λίγο περισσότερο. Τώρα βέβαια είναι 500 εκατομμύρια καταναλωτές στην Ευρώπη. Είναι δύσκολο να έχουμε πληροφορίες που να αφορούν τον καθένα ξεχωριστά. Κάτι άλλο μου φαίνεται, που μου φαίνεται σημαντικό, γιατί είμαι και εισηγητή για την εκδομοδότηση της Επιτροπής Γεωργίας, είναι λαμβάνοντας υπόψη ε, τα όσα λέμε εδώ στο Κοινοβούλιο, υπάρχει και η, αλλαγή του κλίματος, η άνοδος της θερμοκρασίας στον πλανήτη μας. Επομένως, θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, όχι μόνο για τα τρόφιμα, ας πούμε, αυτά καθεαυτά και τη συντήρηση των τροφίμων, αλλά όταν έχουμε ένα τρόφιμο, το οποίο είναι ζωικής προέλευσης και αυτό το ζώο, ας πούμε, αυτό το προϊόν μάλλον φτάνεται στο Βέλγιο. Έχει γεννηθεί στον Καναδά, έχει μεγαλώσει στην Αυστραλία και καταλήγει το επεξεργασμένο προϊόν εδώ στο σούπερ μάρκετ στο Βέλγιο. Ε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το ζώο αυτό έχει κυκλοφορήσει, έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. Και όλα αυτά επηρεάζουν και την αλλαγή του κλίματος και, κάπου θα πρέπει αυτό να αναφέρεται αυτή η πληροφορία τέλο πάντων, με πολύ, η πληροφορία δηλαδή της προέλευσης, που γεννήθηκε, που μεγάλωσε, γιατί στο μέλλον θα είναι απαράδεκτο να χρησιμοποιούμε και να καταναλώνουμε τέτοιου είδους ε, προϊόντα, ε, τα οποία έχουν ταξιδέψει ε, εκατοντάδες χιλιόμετρα για να φτάσουν. Τέλος πάντων, υπάρχουν πολλές πληροφορίες που θα πρέπει να καταλήξουν στον καταναλωτή για να μπορεί και αυτός, ε, έχοντας πλήρη γνώση των όσων συμβαίνουν, να μπορεί να επιλέξει. Τέλος πάντων, συνοψίζω λέγοντας ότι πρέπει να είμαστε απλοί. Να δίνουμε μονάχα τις πλέον απαραίτητες πληροφορίες. Αυτό είναι, αυτός είναι ο στόχος μας εδώ. την αποστολή μας εδώ. Uh, um, Ευχαριστώ, κυρία Παρβανόβα. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς, νομίζω ότι για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό τα πράγματα να παραμείνουν απλά και φιλικά προς τον καταναλωτή. Διότι τώρα συζητάμε τι να βάλουμε μπροστά στην ετικέτα, τι να βάλουμε πίσω από την ετικέτα και μπορεί να καταλήξουμε με μια νομοθεσία η οποία θα προτείνει να έχουμε ένα ολόκληρο φυλάδιο μισού μέτρου για ένα μικρό κουτάκι σοκολάτα. Είναι απαραίτητο για το μέσο καταναλωτή να έχει πληροφορίες οι οποίες είναι απαραίτητες για πανεπιστημιακού επίπεδου αναλυτές χημίας. Και τι σκοπό εξυπηρετούν αυτές οι πληροφορίες. Νομίζω ότι μπορούμε κάλλιστα να συνδυάσουμε το θέμα του GTA με ένα φανάρι, να έχουμε ένα πράσινο, κόκκινο και πορτοκαλί σήμα, το οποίο θα μας δείχνει λίγο τι περιεκτικότητα έχουμε σε λίπη, σε σάχαρα και σε ενέργεια. Αυτά ενδιαφέρουν τον καταναλωτή. Αυτά θα μπορούσε να είναι μπροστά στην ετικέτα του πακέτου της συσκευασία και από εκεί και πέρα λεπτομέρειες μπορεί να υπάρχουν στο πίστιο τμήμα, αλλά φαντάζεστε τώρα να έχουμε ενδελεχείς πληροφορίες για τη χώρα προέλευσης το κατά πόσον θα αρέσει στους καταναλωτές ε, το μοσχάρι από την ε, ε, Αργεντινή από ότι το μοσχάρι από τη Βουλγαρία και ε, συγγνώμη που το λέω αυτό, υπάρχουν και ντομάτες που είναι σαν πλαστικές ε, σε αντίστοιχη με αυτές που παράγονται φρέσκες σε άλλες χώρες. Υπάρχει το θέμα της χώρας προέλευσης βέβαια, είναι πάρα πολύ σημαντικό, θεωρείται προτεραιότητα για τις επιλογές τους, αλλά ακολουθούν και τις τιμές, ακολουθούν και τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται ένα προϊόν, ε, αλλά πρέπει οι οδηγίε που θα του δίνουμε να είναι απλέ, περιεκτικές. Υπάρχουν πανεπιστήμια τα οποία γνωρίζω, κυρίως στην ε, Ολλανδία, που ασχολούνται με το θέμα της ε, πληρότητα των πληροφοριών. Υπάρχει μια ολόκληρη επιστήμη πίσω από αυτό, τι θα βρίσκεται στι συστάσει, τι θα βρίσκεται στο φυλάδιο ή οτιδήποτε άλλο, το οποίο θα στοχεύει στον καταναλωτή και στον ευρύτερο πληθυσμό και νομίζω ότι θα πρέπει να λάβουμε και συμβουλές από κάποιον εμπειρογνώμονα και να δούμε τι γίνεται με όλες αυτές τις 290 ή δεν ξέρω πόσες είναι αυτές οι τροπολογίες, διότι δεν είναι τη εμπειρογνωμοσύνη αυτή τη επιτροπή να αποφασίσει τι είναι καλό και τι είναι κακό, γιατί όπω ξέρετε έχουμε και πάρα πολλέ ομάδε πίεση ε, πίσω μα. Ευχαριστώ. Ο κύριο Φαμπ. Και μετά η κυρία Γκέπχαρτ. Και τέλο ο κύριο Μωτή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος γιατί συμφωνώ με το περιεχόμενο σε αυτά που είπε η κυρία Βάισμπεργκερ σε γενικές γραμμές εφόσον η κυρία Σάλντε Μόζερ ξεκινά ένα νέο ξεκίνημα σε αυτό το φάκελο για την Επιτροπή μας, θα ήθελα να ε, ε, την ευχαριστήσω για τις προτάσεις της που μας διευκολύνουν να επιτύχουμε το στόχο μας, δηλαδή να γνωρίζουμε ποιες ε, είναι οι διατροφικές αξίες των στοιχείων που τρώμε ε, επίσης η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς μέχρι στιγμής είχε συμμετάσχει στις συζητήσεις αυτές μόνο για γνωμοδότηση και γι' αυτό αναρωτιέμαι αν σύμφωνα με το άρθρο 59 δεν θα μπορούσε ο φάκελος αυτός να να ε, περιληφθεί σαν ένα μέτρο για την εσωτερική αγορά και την προστασία του καταναλωτή διότι εδώ πρόκειται ουσιαστικά ε, για πληροφορίες που είναι φύσεως εσωτερικής αγοράς και προστασίας του καταναλωτή ε, Ο ελέγχθη ότι ο Τσέρτσιλ ε, πίστευε τις, ε, ε, τις στατιστικές τις οποίες μόνο αυτός είχε καταρτήσει. Οπότε δεν ξέρω τι επιθυμούν οι καταναλωτές τώρα. Θέλουν να καταλάβουν πιο εύκολα την ποικιλία των τροφίμων χωρίς να χρειαστεί να πληρώσουν πολύ ακριβά για αυτήν την ποικιλία ή ε, θέλει ο καθένας να ξέρει ακριβώς τι τρώει από κάθε κατηγορία οπότε χρειαζόμαστε ίσως ένα κόκκινο φωτάκι, μια προειδοποίηση ε, οπότε πρέπει να δούμε τι κάνουν ορισμένοι ε, παραγωγοί ή ε, και αν αυτές οι πληροφορίες μας ικανοποιούν ή χρειάζεται κάτι παραπάνω οπότε να αξιολογήσουμε αν επαρκούν οι πληροφορίες που δίδονται και αν μην χρειαστούν τόσες τροπολογίες όσο στην προηγούμενη φορά. Η κυρία Γκέπχαρτ Θέλω να ευχαριστήσω την Κριστίν Μόζερ για την καλή δουλειά που έκανε και θα ήθελα εδώ να ε, επιβεβαιώσω αυτά τα οποία είπε. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο, ε, ε, με τον οποίον προχώρησε στην βελτίωση της εκθέσεως Βερνιό διότι αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να καταλάβουν τίποτα οι νέοι ευρωβουλευτές. Ορισμένα σημεία πρέπει να διευκρινιστούν, διότι τότε δεν θα καταρτίζαμε μία νέα έκθεση, αλλά πρέπει να είμαστε επιλεκτικοί στα σημεία τα οποία θα επαναλάβουμε και να επαναλαμβάνουμε μόνο ότι είναι αναγκαίο για να μην χρειαστούμε στο τέλος πάλι 200-300 τροπολογίες για να καταλήξουμε στους ίδιους συμβιβασμούς που καταλήξαμε και την προηγούμενη φορά. Εγώ ήθελα να επανέλθω σε μια παρατήρηση της κυρίας Βάισμπεργκερ και ίσως θα ήταν καλό και η Κρίστερ θα μπορούσε να το πράξει να μας εξηγήσει τι εννοεί με αυτή την επισήμανση διότι ίσως υπάρχουν παρανοήσεις. Εγώ νόμιζα ότι ορισμένοι ε, ήθελαν ε, να, υπάρχει μία επισήμανση ε, με τρία φωτάκια κόκκινο, κίτρινο και πράσινο και θα λέει που κατατάσσεται κάθε προϊόν. Δεν εννοούμε αυτό στην επισήμανση. Εμείς εννοούμε ε, να αναφέρονται ε, τα συστατικά και να λέγεται υπάρχει πολύ ζάχαρη ή λίγη ζάχαρη, πολύ λίπος ή λίγο λίπος. Αυτό είναι ε, μία λύση της επισημάνσεως η οποία είναι πληροφοριακή και αν είναι κάτι καλό θα είναι πράσινο το σήμα και αν είναι κάτι κακό, λίπος παραδείγματος χάρη, κόκκινο ή αντίστοιχα με τη ζάχαρη, ε, διότι ίσως αυτό θα ήταν μια καλή λύση και θα έπρεπε ίσως Κρίστελ εσύ ή κάποιος άλλος να διευκρινίσει ότι εδώ ε, προσπαθούμε να κάνουμε κάτι λογικό και όχι απλώς ε, επειδή ορισμένοι έχουν μία λαθασμένη εικόνα του τι γίνεται θα απορρίψουμε τη συνολική ιδέα. Αυτές είναι οι πληροφορίες οι οποίες όντως μπορεί να είναι χρήσιμες στον καταναλωτή. Ευχαριστώ. Κύριε Γκέπχαρτ. Το κόκκινο σημαίνει μην οδηγείτε. Σημαίνει επίσης και μην λέτε ψέματα. Διερωτώ με. Ο κύριος Μότι. Το, οι σοσιαλιστές έχουν το κόκκινο, άρα το κόκκινο είναι ωραίο χρώμα και όχι μόνο απαγορευτικό. <laughs> είναι τόσο ωραίο. Do we have Mr. Motti here? Ο κύριος Μότι, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πρέπει να πω ότι με προλάβατε ήθελα να εκφράσω την προσωπική μου άποψη, όχι για την έκθεση, την οποία παραδέχομαι ότι δεν έχω διαβάσει, αλλά για τα όσα άκουσα εδώ στη συζήτηση, την οποία παρακολούθησα. Το φανάρι θα μπορούσε να δίνει την εντύπωση στον καταναλωτή ότι βρίσκεται ενώπιον μιας επιλογής. Και επειδή εμείς είμαστε συνηθισμένοι να προχωράμε με το πράσινο και να σταματάμε με το κόκκινο, θα ήθελα να εκφράσω μια ε, αντίρρηση για μια ετικέτα η οποία ουσιαστικά θα περιλαμβάνει μία ένδειξη η οποία θεωρείται εκ των προτέρων ως μία ένδειξη συμπεριφοράς που πρέπει να ακολουθείτε. Τέλος πάντων αυτή είναι μία προσωπική απορία. Θεωρώ ότι το περιεχόμενο της ετικέτας θα πρέπει ούτως ή άλλως να είναι βανάγνωστο για τον ε, καταναλωτή. Διότι αν εμείς θέλουμε να δώσουμε πραγματικά πληρέστατες πληροφορίες, θα πρέπει να πούμε ακόμα και αν τα σάκχαρα που ε, περιλαμβάνονται σε ένα μεταποιημένο προϊόν είναι σακχαρόζι, γλυκόζι ή κάτι άλλο. Γιατί, για παράδειγμα, για ένα διαβητικό είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει το γλυκαιμικό δίκτυο αυτού που καταναλώνει και η ζάχαρη δεν είναι πάντα το ίδιο. Και η ινσουλίνη έχει διαφορές, διαφορετικές επιπτώσεις ανάλογα με τη ζάχαρη που καταναλώνεται. Να πω μια προσωπική γνώμη, δεν έχω διαβάσει την έκθεση, οπότε μπορεί να λέω πράγματα τα οποία έχουν ήδη επαναληφθεί και έχουν προβλεφθεί. Πρόκειται για ένα μεταποιημένο προϊόν και επίσης έχουμε και ένα προϊόν το οποίο μπορεί να έχει διαιτητικά χαρακτηριστικά. Τοποθετείται δηλαδή στην αγορά και απευθύνεται σε καταναλωτές που ενδιαφέρονται ιδιαίτερα ε, σε σχέση με τις διατροφικά χαρακτηριστικά με το προϊόν. Σε αυτή την περίπτωση ή θα πρέπει να έχουμε υποχρεωτική ή ε, κατ' επιλογή νομοθεσία, αλλά θα πρέπει να υποδεικνύονται μία σειρά από επιπρόσθετα στοιχεία. Διότι ο καταναλωτής αυτή τη μορφής είναι ιδιαίτερα προσεκτικός σε τέτοια θέματα. Ο μέσος καταναλωτής μπορεί απλά να θέλει να ξέρει αν τρώει ένα τρόφιμα που έχει πολλά λιπαρά, πάρα πολλά λιπαρά γιατί αυτό που κοιτάμε είναι κυρίω τα λιπαρά σήμερα και αφορά τη διατροφή μα ή ποια είναι η εξισορρόπηση των βασικών στοιχείων και αυτό θα μπορούσε κάλλιστα να παρουσιάζεται με μία απλή ετικέτα και σε αυτό είμαι υπέρ του GDA το οποίο αναφέραμε. Μία τελευταία πολύ γρήγορη παρατήρηση για το χώρο προέλευσης ή το χώρο μεταποίησης των προϊόντων. Ε, όσον αφορά στην Ιταλία, εγώ γνωρίζω ότι επί του παρόντος το γάλα που καταναλώνω ο χώρος στον οποίο παστεριώθηκε το γάλα αναφέρεται μόνο στις συσκευασίε ε, φρέσκου γάλακτος, αυτό δηλαδή που λύγει πολύ σύντομα. Ενώ στο μακράς διαρκείας γάλα δεν είναι υποχρεωτική αυτή η αναφορά. θεωρώ ότι είναι δικαίωμα του καταναλωτή να γνωρίζει αν το γάλα το οποίο πίνει, το οποίο μπορεί στην ε, ε, συσκευασία να έχει μια τεράστια ε, μάρκα ε, της ε, χώρας, της πόλης στην οποία ζει και εκεί αυτή είναι η τάση να παίρνουμε γάλα το οποίο θεωρεί ότι παστεριώνεται στην πόλη του θα πρέπει να γνωρίζω ίσως αν είναι από κάποια άλλη χώρα το αν έρχεται από κάποια άλλη χώρα βέβαια δεν σημαίνει απαραίτητα ότι δεν είναι καλή ποιότητα, αλλά θεωρώ ότι αυτή η πληροφορία θα πρέπει να αναγράφεται στη συσκευασία Ευχαριστώ πολύ κύριε Μότι Τώρα πριν δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον κύριο Γκουδελάια, τον εκπρόσωπο, η κυρία äh, Ευχαριστώ. Ήθελα να αναφερθώ στο σχόλιο της κυρίας Γκέρμπερ. Κατάλαβα αυτό, αυτή την επισήμανση, ε, αλλά υπάρχει μία συνολική και μία καταπερίπτωση ε, Είναι οι προτάσεις οι οποίες υπάρχουν. Για ένα προϊόν υπάρχει μία επισήμανση και συμφωνώ μαζί σας αυτό. Αλλά εγώ είμαι ε, ενάντια στις χρωματικές κατατάξεις των, των διαφορετικών θεματων ε, θεμάτων. Δηλαδή, εάν ε, ε, είχαμε μία διαβάθμιση κόκκινο-κίτρινο-πράσινο για τη ζάχαρη παραδείγματος χάρη, δεν συμφωνώ διότι ενδέχεται να υπάρχει ένα κόκκινο για μία διατροφική τιμή που θα αποτρέψει κάποιον από πότε θα ισχύσει αυτό δηλαδή πού θέτουμε το όριο, τι θα πάει στα κόκκινα ή στα κίτρινα και ε, γι' αυτό προβληματίζουμε διότι θα πρέπει να συγκεντρώσουμε τις πληροφορίες πολιτικά δηλαδή εάν κάποιος δέχεται ή όχι αυτές τις καθημερινές διατροφικές τιμές και τα GDA και δίνουμε στον, ε, ε, στον καταναλωτή τη δυνατότητα να επιλέξει τι τρώει κάθε μέρα σε σχέση με τις διατροφικές δικές ανάγκες ε, ανά ημέρα. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ε, τι θα γίνει με αυτές τις διατροφικές πληροφορίες. Παραδείγματο χάρη έχουμε το συνάδελφο ή στην Επιτροπή Γεωργίας, δεν ξέρω το όνομά του, ο οποίος είπε ότι όσον αφορά τα GDA θα πρέπει να αναφέρονται στις μέσες τιμές. Είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να πει κανείς ε, ε, πρέπει να είναι μέσες τιμές, αλλά εγώ θέλω να έχω ένα σημείο Δηλαδή σαν γυναίκα δεν έχω τις ίδιες τιμές με τους άντρες. Εάν είμαι πιο νέα μπορεί ε, οι ανάγκες μου να είναι χαμηλότερες και ε, βλέπω ότι στην Αμερική είναι πολύ πιο ακριβές. Υπάρχει δηλαδή ε, ένα κουτί που λέει Nutritional Facts, Daily Value. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτή είναι η καλύτερη ενημέρωση του καταναλωτή που είναι, ε, ε, είναι πληροφόρηση ούτε προτροπή ούτε αποτροπή. Ευχαριστώ και τώρα έχουμε τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κατόπιν η κυρία Σαλτεμόζε θα ολοκληρώσει. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Βαγνιό, η οποία είχε προετοιμάσει την έκθεση αυτή στην προηγούμενη θητεία. Ε, προφανώς θα συνεργαστούμε τώρα ε, και μαζί σας ε, με την κυρία Σάλτερ Μόζερ για να δούμε τι μπορούμε να προχωρήσουμε, τι μπορούμε να κάνουμε. Να σχολιάσω λίγο αυτά τα οποία ακούστηκαν, κυρίως για τις προτινόμενες μερίσιες προσλήψεις. Ε, έχουν υπολογιστεί με βάση τις ανάγκες του μέσου ατόμου, τέλο πάντων, για να δώσουμε μια κατευθυντήρια γραμμή για το τι πρέπει να καταναλώνει ο καθένας δεν έχουμε πρόθεση να ενημερώσουμε και να εκπαιδεύσουμε τον καταναλωτή τι πρέπει να κάνει. Χρειάζεται και άλλες προφορίες ο καταναλωτής ε, για το τι πρέπει να τρώει και πόσο. Απλώς ε, οι, οι, οι πληροφορίες αυτές που τώρα πάνω στην ετικέτα ε, θα του δώσουν κάποιες συμπληρωματικές πληροφορίες όσον αφορά τις ημερήσιες προσλήψεις. Ένα αυτό. Δεύτερον, με τα φανάρια, κόκκινο, πράσινο κτλ. Σας υπενθυμίζω ότι δεν έχουμε προτείνει να εφαρμόσουμε αυτά τα, αυτό το μέτρο του φαναριού, του κόκκινου, του πράσινου και του πορτοκαλί. Ε, κάθε κράτο μέλο θα πρέπει να εφαρμόσει ένα σύστημα το οποίο να βολεύει καλύτερα του καταναλωτές ε, που είναι ανάλογα με τις παραδόσεις του κράτου, με τι συνήθειε του κράτου. Ε, γι' αυτό δεν επιβάλλουμε κάποιο σύστημα. Είπαμε κάθε κράτο μέλο, ανάλογα με την ιστορία του να μπορεί να δημιουργήσει ένα σύστημα, ένα σύστημα το οποίο να μπορεί να αναγνωριστεί και από του άλλου, αλλά και που να ενημερώνει σωστά του καταναλωτέ, Να είναι ένα στέρι, να είναι ένα κλειδί, να είναι ένα ε, ε, φανάρι κόκκινο, πράσινο κτλ. Δικαίωμα κάθε κράτους μέλους να εφαρμόσει το δικό του σύστημα. Τώρα, εάν σαν, αν σε ένα κράτος μέλος υπάρχει μια προϊστορία σχετικά με τα κόκκινα φανάρια τέλος πάντων, ε, γιατί οι αρχές οι, οι καταναλωτών ή δεν ξέρω εγώ τι διανομής έχουν εφαρμόσει αυτό το σύστημα με τα διάφορα χρώματα κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί, α το εφαρμόσουν και α ενημερώσουν και τα άλλα κράτη-μέλη για να, μπορεί να, είναι, να μπορούν να καταλαβαίνουν και οι καταναλωτέ σε άλλα, κρατο, άλλα κράτη-μέλη τι συμβαίνει. Τώρα, ο κατάλογο των συστατικών. Ε, είναι μεγάλο το θέμα και όπως και η προέλευση. Δεν θελήσαμε να επιβάλλουμε ένα υποχρεωτικό σύστημα. Το σύστημα είναι προαιρετικό αρκεί βέβαια να μην ε, ε, κοροϊδεύουμε τον καταναλωτή. Και όταν έχουμε να κάνουμε με μεταποιημένα προϊόντα, παραδείγματος πίτσα, τελευταία επεξεργασία ε, μετράει. Έστω και αν το επιμέρους, ε, τα επιμέρους συστατικά προέρχονται από διάφορες χώρες ε, του κόσμου. Ας πούμε, η, η, η ντομάτα της πίτσας μπορεί να προέρχεται την Κίνα, δυστυχώς. Και λέω δυστυχώς διότι στην Ευρώπη παράγουμε πολλές, πολλές ντομάτες. Αλλά τέλος πάντων. Πολλοί λένε ότι δεν θα πρέπει να ε, μεταφέρουμε, να, να εισάγουμε ντομάτες από τη, την άλλη άκρη του κόσμου. Τέλος πάντων, ένα άλλο στοιχείο το οποίο πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι δεν ε, ρυθμίζουμε μέσω αυτό, αυτού του σχεδίου κανονισμού τα διαιτητικά προϊόντα, τα διαιτητικά τρόφιμα. Αυτό είναι ξεχωριστό κείμενο. Εδώ μιλάμε για τρόφιμα παραδοσιακά, ας πούμε, που απευθύνονται στο ευρύ κοινό. Και αυτή είναι και η δυσκολία μας, γιατί το ευρύ κοινό, ξέρετε, ότι αφορά τα παιδιά, τους αλλεργικούς, τους διαβητικούς, τους ηλικιωμένους, τους ενήλικες που αθλούνται πολύ. Επομένως θα πρέπει μέσω αυτής της επισήμανσης, μέσω των, ε, της ετικετοθεσίας, ε, τα κάποια στοιχεία όπως το αλάτι, τα κορεσμένα, τα κόριστα κτλ, ε, μέσω των, ποσοστό, των ποσοστών προτινόμενης ημερήσης πρόοδος κτλ, μέσω όλων αυτών των στοιχείων θα πρέπει όλοι να ενημερώνονται και να κάνουν μια πεφωτισμένη επιλογή. Βέβαια, κανείς δεν έθιξε αυτό το θέμα, διότι ίσως να υπάρχει ομοφωνία, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο μας ε, απασχολεί, είναι το μέγεθος ε, των γραμμάτων, των στοιχείων ε, και σε αυτό υπάρχει μια συζήτηση. Πρέπει το μέγεθος των γραμμάτων να είναι τέτοιο έτσι ώστε να μπορεί να το διαβάσει κανείς στα, στα, στα μπουκάλια αυτά εδώ, πούμε, για παράδειγμα, λίγοι καταφέρνουν να διαβάσουν ε, τι γράφει. Λοιπόν, είναι μπλε, πάνω στο μπλε. Το νερό μέσα είναι μπλε, τι να διαβάσει ο άλλος. Επομένως, θα πρέπει ακριβώς ε, μέσω της πρότασής μας να έχουμε μία επισήμανση η οποία να μην πιάνει μένει και πολύ χώρο, να στο ε, να μοιράζεται στο μπροστινό και στο πίσω μέρος της συσκευασία, ε, όταν έχουμε να κάνουμε με μια τετράγωνη, ένα κουτί τέλος πάντων και όχι ένα μπουκάλι και θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίε για τους καταναλωτές. Αυτά με λίγα λόγια. Αυτές είναι οι προτάσεις μας ε, για την συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Σάλντο Μόζερ. Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας. Νομίζω ότι αυτό αποδεικνύει ότι δεν είναι απαραίτητο να είναι πανεύκολο να βρούμε μια λύση. Υπάρχουν πάρα πολλοί ενδιαφερόμενοι, πολλές ε, απόψεις ερίζουν. Πολλά έχουν να κάνουν με πολιτική και κάποια έχουν να κάνουν και με διαφορετική νοοτροπία και διαφορετικούς πολιτισμούς στα κράτη-μέλη. Είναι πράγματα όμως τα οποία επηρεάζουν και την καθημερινότητά μας. Όταν μιλάμε λοιπόν για τα GDA, θα ήθελα να σας δώσω ένα παράδειγμα, το οποίο νομίζω αποδεικνύει πολύ καλύτερα αυτό που σας έδωσα ως πρώτο παράδειγμα. Αν πάρετε ένα ποτήρι γάλα και ένα ποτήρι κοκακόλα και χρησιμοποιήσετε επισήμανση GDA, όπως προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τότε το αναψυκτικό θα φαίνεται στον καταναλωτή ως κάτι το οποίο είναι πιο υγιεινό από το γάλα, γιατί έχει λιγότερα λιπαρά και επομένως αν είστε καταναλωτής και προσπαθείτε να διαπιστώσετε αν είναι καλό ή κακό, αυτό θα είναι αρνητικό στοιχείο. Και αυτό είναι το επιχείρημα που προσπαθώ να σας περάσω. Δεν πρέπει να παραπλανούμε τον καταναλωτή, πρέπει να τον ενημερώνουμε. Τέλος πάντων, να μην ακολουθήσουμε άλλο αυτή την άγουσα αυτή τη στιγμή. Ακούω και συζητήσεις εδώ εξ αριστερών. Θα ήθελα να ζητήσω λοιπόν από τους κοιόδης εισηγητές να μας κάνουν μια πιο διεξοδική συζήτηση ε, σε σχέση και με την έκθεση που λάβαμε, να δούμε αν υπάρχουν στοιχεία τα οποία θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε ως βάση συμφωνίας, για να μην ξεκινήσουμε εκ του μηδενός, να βρούμε ένα-δύο-τρία θέματα τα οποία θα μπορούσαμε να επεξεργαστούμε περαιτέρω. Επιπλέον, οποιοδήποτε από εσά θέλει, ανα πάσα στιγμή μπορεί να προτείνει τροπολογίες. Να πω τώρα ότι η δική μου η θέση για το πακέτο για τις πληροφορίες για τη διατροφή είναι ότι θα πρέπει ο καταναλωτής να επαφολείται από το θέμα αυτό στο τέλος, ε, διότι ο καταναλωτής είναι αυτός ο οποίος ε, πρέπει να μπορεί να κάνει μια επιλογή και όχι ο έμπορος να πουλήσει το προϊόν του. Αυτός είναι αυτός ο οποίος θα πρέπει να κάνει επιλογή για την καθημερινότητά του και αυτή θα πρέπει να είναι η αρχή που θα πρέπει να διέπει αυτό που θα κάνουμε για την έκθεση. Ευχαριστώ πολύ και προσβλέπω στις συζητήσεις που θα κάνουμε για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ κυρία Σαλντεμόζε, ευχαριστώ και τους ε, συναδέλφους, ευχαριστώ τους εμπειρογνώμονες, τη γραμματεία, τους διερμηνείς. Εγώ πείνασα. Θα συνεχίσουμε το απόγευμα πατατάκια, πίτσα, ντομάτες, γάλα. Καλή όρεξη.